Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχουμε σήμερα μία δημόσια κρόαση αφιερωμένη στην συνεργασία μεταξύ πολιτική, και ε, πολιτικοστρατικής συνεργασίας, ένα θέμα το οποίο επέλεξαν το σύνολο των πολιτικών ομάδων. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημέρηση διάταξη, θα προχωρήσουμε να σας ε, θυμίσω πως μερικές γλώσσες δεν μεταφράζονται σήμερα. Le le, le, le bulgare, le tchèque, le slovaque et l'estonien. Euh, la réunion est Η συνεδρίαση μεταδίδεται απευθείας στο web stream και θα ήθελα, εφόσον δεν έχουμε ξανασυναντηθεί σε αυτό το σχήμα της Υποεπιτροπής εδώ και κάποιες εβδομάδες, πριν να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, να σας θυμίσω ότι με την ευκαιρία αυτή της ε, αεροπορική τραγωδίας που κόστησε, στήχησε τη ζωή σε πολλούς ε, συναδέλφους βουλευτές αλλά και στελέχη των ε, πολωνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Η τραγωδία της 10ης Απριλίου στο Σμόλενγκ, τότε στην υπο... ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής είχα υποβάλει σε όλους τα συλληπιτήριά μας, ε, στους ε, πολωνούς συναδέλφους, πρώτα στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Ζέζι Μπούζεκ, αλλά και στους Πολωνούς ευρωβουλευτές και εθνικούς βουλευτές. Πρόκειται για μια μεγάλη απώλεια για μια χώρα που είναι εξαιρετικά σημαντική για όλες τις εργασίες που κάνουμε για την πολιτική κοινή ε, ασφάλειας και άμυνας. Και ήθελα έτσι να ε, σκεφτούμε για λίγο ε, τους ανθρώπους αυτούς που χάθηκαν και τις οικογένειές τους. Για αύριο υπάρχει μια πιθανότητα αλλαγή στο πρόγραμμα. Είχαμε προβλέψει μια συνεδρίαση για το Κωσυφοπαίδιο με την ε, ε, αποστολή Ελέξη με τον ε, στρατηγό Κέρμαμπο, αλλά μας ενημέρωσε πως είναι πιθανό να αναβάλει την παρουσία του εδώ. Θα σας ενημερώνω. Είμαστε σε επαφή μαζί του. Τώρα, εάν αυτή η ανταλλαγή απόψεων για το κοσμοπέδιο δεν μπορέσει να λάβει χώρα, αυτό που θα σας πρότεινα υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, γιατί γνωρίζετε ότι στις 31 Μαρτίου η, τα μέλη της ε, ΔΕΕ της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης ε, ανακοίνωσαν την έναρξη της διαδικασίας που θέτει πέρα στην Συνθήκη των Βρυξελών καθώς και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ε, ΔΕΕ. Μετά από αυτήν την απόφαση ήθελα να συζητήσουμε στο σχήμα ΣΕΝΤΕ και κλεισμένο των θυρών. Τι συνέπειε θα έχει τέτοιο, κάτι τέτοιο όσον αφορά την διακοινοβουλευτική συνεργασία για θέματα Άμυνα. Θα μπορούσαμε στο τέλο τη ακρόαση να το συζητήσουμε. Οπότε, σε περίπτωση που δεν γίνει η συνεδρίαση για το κοσυφοπαίδιο, θα μπορούσαμε να συνεδριάσουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα θέμα για το οποίο ο συνάδελφο Ντάφ έχει προετοιμάσει ένα έγγραφο, το οποίο ίσω θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. να σας ανακοινώσω πως η επόμενη έκθεση πρωτοβουλίας θα αφορά ακριβώς τη συνεργασία την πολιτικό-στρατιωτική, αυτό το θέμα δηλαδή που θα μας απασχολήσει σήμερα και έχουμε την εγνωμοδότηση της κυρίας Κοπά για τη ζωριφόρους ε, Ε, η έκθεση για την ε, για την ανακοίνωση της Κομισιόν για τα βιοχημικά όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί σε ποια πολιτική ομάδα θα ανατεθεί η έκθεση αυτή. Αυτά λοιπόν για τις ανακοινώσεις και τις μελλοντικέ μας ε, συνεδριάσεις. Σήμερα λοιπόν ομόφωνα αποφασίσαμε το σύνολο δηλαδή των πολιτικών ομάδων εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την ε, διεξαγωγή μιας δημόσιας ακρόσης για το θέμα της πολιτικοστατικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει πολύ σημαντικές διαστάσεις, είναι πολύ επίκαιρο, καταρχήν υπό το φως της συνθήκης της Λισαβόνας, που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, πρέπει να έχει μια τέτοια διπλή διτή προσέγγιση, πολιτική και στρατιωτική, σε όλες ε, τις επιχειρήσεις που γίνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ και επίσης ένα θέμα που είναι ευαίσθητο όσον αφορά τα θέατρα επιχειρήσεων όπως το Αφγανιστάν, για το οποίο έχουμε ήδη εκφράσει θέση, λάβει θέση, αλλά και ένα θέμα το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο και στο ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ ξεκινά την ε, αναθεώρηση των στρατηγικών του δογμάτων και ε, ω εκ τούτου η συζήτηση αυτή είναι όλα ένα και πιο ενδιαφέρουσα. Η πολιτικοστρατηγική συνεργασία στην Ένωση αποτελεί την μεγάλη προστιθέμενη αξία και την μεγάλη πρωτοτυπία της ε, ΚΕΠΑ για να το συζητήσουμε έχουμε προσκαλέσει διάφορους ερευνητές αλλά και πρακτικούς ε, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα δύο πακέτα. Ένα πρώτο κομμάτι το οποίο σχετίζεται περισσότερο με θεσμικά ζητήματα, δηλαδή ποια είναι τα μέσα που έχουν δημιουργηθεί τελευταία και πρόσφατα είχαμε ένα παράδειγμα με την CN5, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού όπου γίνεται ο προγραμματισμός της διαχείρισης των κρίσεων και συμπεριλαμβάνεται η πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τις, ε, την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, να δούμε ποιο σύνδεση θα υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες αυτές υπηρεσίες ε, για τη διαχείριση ε, κρίσεων από πολιτικής και από στρατιωτικής πλευράς και έπειτα θα ζητήσω από τους εμπειρογνώμους να εστιάσουν την προσοχή στη δεύτερη φάση, στα πιο πρακτικά ζητήματα, όπως δηλαδή αυτά παρουσιάζονται επί τόπου, με βάση διάφορες επιχειρήσεις που έχουν ήδη γίνει. Για το πρώτο κομμάτι λοιπόν θα έχουμε τέσσερις ομιλητές, στους οποίους ε, θα ζητήσω να μιλήσουν για ένα δεκάλεπτο, ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε τον κύριο Didier Lenoir, που είναι προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, της ΣΕΜΠΕΝΤΕ, τον κύριο Κιόχαν, ε, πάντα δυσκολεύομαι το όνομά του, που είναι επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτο Μελετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ασφαλεία στο Παρίσι, τον κύριο Γκέρεν, που είναι αναπληρωτή διευθυντή Πολιτική στο Κέντρο Διεθνού Συνεργασία του Πανεπιστημίου τη Νέα Υόρκη και με τον κύριο Μάλεγκ που μόλι έχει συντάξει μια μελέτη την οποία του ανέθεσε το Ευρωκοινοβούλιο που ονομάζεται, ονομάζεται τη δημιουργία μια πολιτικοστρατηγική συνεργασία τη ΕΕ και ο αντίκτυπος της συνθήκης της Λισαβόνας. Να σας παρουσιάσω και τους ομιλητές του δεύτερου τμήματος που είναι το πιο επιχειρησιακό. Έχουμε τον κύριο Έρχαρτ που είναι προϊστάμενος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μελετών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια του Ινστιτούτου Ερευνών του Αμβούργου. Το κύριο Ρίτσενς της Ακαδημίας Άμυνας των Κάτω Χωρών η κυρία Φρανσουάζ Κρίλ, που είναι προϊστάμενο τη Επιτροπής τη Διεθνού Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και τον κύριο Ράιτ, που θα έρθει νομίζω λίγο αργότερα, και που είναι διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκινούμε με το πρώτο τμήμα. Διδιέ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι προϊστάμενο τη Υπηρεσία ε, Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού στο εντός της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η διεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε στι αρχές του χρόνου και δεν έχει ακόμα ε, φτάσει στην πλήρη επιχειρησιακή της ε, δυνατότητα. Είμαστε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο και άρα οι δομέ τη ΕΜΠΕΝΤΕ θα κληθούν ακόμη να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Η ομάδα της οποίας ηγούμε αποτελείται από 30 άτομα, τα οποία ε, βασικά προέρχονται από το κύτταρο το πολιτικό στρατητικό που υπήρχε ανέκαθεν στο Συμβούλιο την πρώην διεύθυνση που είχε αναλάβει τη διαχείριση κρίσεων και την πρώην διεύθυνση ε, που ασχολείται με την πολιτική διαχείριση των κρίσεων. Επίσης έχουμε προβλέψει μέσα στο πλαίσιο των υπαλλήλων της διεύθυνσης μια μονάδα στρατηγικού σχεδιασμού η οποία συμπεριλαμβάνει ε, κάποιους εκπροσώπους της Κομισιόν για λόγους προφανής για να διασφαλιστεί δηλαδή η σύνδεση ανάμεσα στις δραστηριότητες που διεξάγει η Κομισιόν και τις δραστηριότητες ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων στον αφορά τη διαχείριση των κρίσεων. Αυτό η ομάδα ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού οργανώνεται σε διάφορες γεωγραφικά τμήματα. Γιατί επιλέξαμε αυτό το πρότυπο αντί για κάποιο άλλο ακριβώς για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση ανάμεσα στην πολιτικοστρατιωτική, πολιτικό και στρατιωτικό σκέλος, γιατί κρίναμε ότι ήταν πιο φρόνιμο να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους ε, υπηρεσία και ότι το να δημιουργήσουμε γεωγραφικά τμήματα θα μας επέτρεπε να εξασφαλίσουμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ήταν αντικείμενο της δημιουργίας της ίδιας της διεύθυνσης να σας πω ότι αυτή η διεύθυνση είναι το αποτέλεσμα εργασιών που ξεκίνησαν υπό την Γαλλική Προεδρία, αλλά την ιδέα την έχουμε επεξεργαστεί εδώ και πιο πολλά χρόνια. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε τη διαδικασία post μετά τον, τον και τον Ε, προτάθηκε καταρχήν στο Hampton Court, μετά από, δηλαδή από εκείνη την ε, διάσκεψη κορυφής του Συμβουλίου. Βασική, μία μάλλον από τις ιδέες είναι ότι η, μια μονάδα διαχείρισης χρήσεων δεν είναι ε, η ίδια αυτός σκοπό, εξυπηρετεί πολιτικούς σκοπού, τους οποίους καθορίζουν οι πολιτικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν και τον πολιτικό έλεγχο και την στρατηγική διαχείριση της διεύθυνσης διαχείρισης κρίσεων. Πρώτη βασική ιδέα και προτεραιότητα είναι ακριβώς ο πολιτικός έλεγχος στις δραστηριότητε ελέγχου, μάλλον διαχείρισης κρίσεων. Και ακριβώς αυτόν τον έλεγχο θέλει να ασκήσει η δική μας διεύθυνση από πλευρά του Συμβουλίου. Αυτός ο πολιτικός στόχος τώρα κάθε φορά δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μέσα διαχείρισης κρίσεων. Ε, οι αποστολέ διαχείριση κρίσεων έχουν λοιπόν ω εντολή να ενταχθούν μέσα σε μια γενικότερη και ευρύτερη προσπάθεια που κινητοποιεί το σύνολο των μέσων, των πόρων, των δυνατοτήτων και τη ενέργεια Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να επιτύχει τον πολιτικό τη στόχο. Αυτές οι δύο διαπιστώσεις δεν ε, είναι επαναστατικές, έτσι λειτουργούν όλα μας τα κρατημέλη και έτσι λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή είναι βέβαια κάπως πιο περίπλοκη. Γιατί βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες της πραγματικής ζωής και τους περιορισμούς που πρέπει κανείς να σεβαστεί. Οι δύο βασικοί περιορισμοί, κατά την άποψή μου, είναι η ανάγκη να, σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση και γιατί πρέπει οπωσδήποτε να, σκεφτούμε, να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες των εργαλείων, γιατί αυτό έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά τους. Μια αστυνομική υποαποστολή δεν θα δώσει πλήρη ικανοποίηση παρά αν σχεδιαστεί και διεξαχθεί σύμφωνα με τις αντιλήψεις της αστυνομικέ ένα δόγμα το οποίο έχει θεσπιστεί με βάση την πείρα που δύσκολα έχει αποκτηθεί. Άρα λοιπόν σεβασμό στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, ανάγκη να σεβαστούμε δηλαδή τη διαδικασία σχεδιασμού, τον τρόπο με τον οποίο το διαχειριζόμαστε και δεύτερος περιορισμός είναι το να διατηρηθεί ένας συνολικός, μια συνολική συνοχή και ένα συγκεκριμένο πολιτικός στόχος. Πώς μπορούμε λοιπόν να λύσουμε αυτήν την εξίσωση. Οι αρμόδιοι θεώρησαν ότι έπρεπε να γίνει διάκριση μεταξύ δύο επιπέδων, του στρατηγικού που είναι αυτό στο οποίο ανήκει το ΣΕΜ5, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού, και ένα δεύτερο επίπεδο, δηλαδή την ολοκλήρωση. Δηλαδή, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα μέσα διαχείρισης κρίσεων, ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι τους, ποια πρέπει να είναι το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο χρησιμοποιούμε Πώς διασφαλίζεται ο συντονισμός όλων αυτών των δραστηριοτήτων, εν πάση περιπτώσει να οριστεί το γενικό πλαίσιο της χρήση των ε, εργαλείων διαχείρισης κρίσεων. Η λέξη κλειδί είναι λοιπόν η λέξη ολοκλήρωση. Στο επιχειρησιακό επίπεδο η λέξη κλειδί δεν είναι τόσο η ολοκλήρωση όσο η συνεργασία. Γιατί ε, να εισάγουμε μια τέτοια διάκριση ακριβώς για να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα του πολιτικού ή του στρατιωτικού εργαλείου ή των εργαλείων όποια και είναι αυτά, να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητά τους ώστε να εξασφαλίσουμε την αποδοτικότητά τους. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, στο στρατηγικό επίπεδο θα ήθελα να πω πιο συγκεκριμένα τι σημαίνουν όλα αυτά σημαίνουν τρεις, ε, τρεις πτυχές. Καταρχήν, ολοκλήρωση των πτυχών των πολιτικών και των στρατιωτικών σε ένα συνεκτικό σύνολο και να διασφαλίσουμε και την συμβολή τους όπως αυτή αναμένεται για την επίλυση κάποιες συγκεκριμένε κρίσεις. Δεύτερος στόχος, ε, να εξασφαλίσουμε αυτή την ολοκλήρωση σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο ορίζουν οι νόμιμες Πολιτικέ αρχές. Και τρίτο στόχος, το να διασφαλιστεί στενή συνεργασία με τα άλλα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους που έχει θέσει. Ο ρόλος της διεύθυνσής μας ποιος είναι, γιατί έλεγα ότι αυτό το στρατηγικό επίπεδο είναι αυτό στο οποίο τοποθετείται η διεύθυνσή μας Θέλουμε να προτείνουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείριση κρίσεων με βάση αυτό που λέμε ε, σύμφωνα με τα μοντέλα της ε, διαχείρισης των χρήσεων, να προετοιμάσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου σε σχέση με τη δέσμευση της Ένωσης και να εξασφαλίσει και τη συνεργασία με τα, τους άλλους φορείς, που παράλληλα με τα φορείς διαχείρισης κρίσεων μπορεί να συμβάλλουν και στην επίλυση της κρίσης. Όσον αφορά το επιχειρησιακό επίπεδο, θα μιλήσω σύντομα μόνο γιατί είναι τμήμα του επόμενου πάνελ, να υπογραμμίσω μόνο δύο-τρία στοιχεία. Ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω ότι μια προϋπόθεση εκ των όνων ε, ε, για την, για την συγκεκριμένη διεύθυνση είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί να είναι ε, αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα του κάθε μέσου. Δεύτερον, να επιμείνουμε για το γεγονός ότι ο σεβασμός στην ιδιαιτερότητα δεν ε, πρέπει να θεωρηθεί ως μια απόλυτη βούληση για ανεξαρτησία. Όχι, πρέπει να υπάρχει στενός συντονισμός Και να υπογραμμίσουμε επίσης ότι δεν είναι κάτι τελείως νέο. Έχουμε ήδη ε, πειραματιστεί πάνω σε αυτή τη συνεργασία στην ε, επιχείρηση Ταλάντα, στην επιχείρηση UNFOR Η συνεργασία αυτή λοιπόν μέσα στο σεβασμό της διαφοράς λειτουργεί. Τι χρειάζεται τώρα για να λειτουργήσει σε επιχειρησιακό επίπεδο αυτή η συνεργασία, να έχουμε καθορίσει τρόπο συνεργασίας επιτόπου και αυτός είναι ένας από τους στόχους ε, του μοντέλου διαχείρισης των κρίσεων. Έπειτα χρειάζονται φορείς που έχουν την συνήθεια να συνεργάζονται. Μιλώ εδώ για τους υπευθύνου για τα στρατηγία των, των, των επιχειρήσεων, δηλαδή που γνωρίζουν τις διαδικασίες επίσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης και που θα αποτελούν ένα σύνολο σαφές, ξεκάθαρο όσον αφορά τις ευθύνε του καθενός. cette, cette dichotomie να σας ε, να υπογραμμίσω ότι η διάκριση που, που ανέφερα ανάμεσα στην στρατηγική, στο στρατηγικό σχεδιασμό και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι είναι κάτι που οδηγεί σε ε, ε, διάκριση των δύο διαδικασιών. Δηλαδή υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ όλων αυτών, ε, από το ένα περνάμε στο άλλο. Ε, το, σήμερα όλες οι κρίσεις έχουν ε, από... Ε, έχουν μάλλον πολιτικές, πολιτικά στοιχεία αλλά και επιχειρησιακά και άρα κάθε πολιτική δράση μπορεί να έχει επιπτώσεις επιτόπου. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει μια ε, ε, αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ε, πολιτικές και επιχειρησιακές πτυχές του σχεδιασμού. Για την πολιτικοστατική συνεργασία, λοιπόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει προεγνήσια βούληση να προχωρήσουμε, να εμβαθύνουμε διαρκώ αυτή τη διάσταση στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημιουργία του ΣΕΜ5, τη Διεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Σχεδιασμού, είναι μια απόδειξη γι' αυτό. Είδα ότι τα έγγραφά μας αποτελούν βιβλιογραφία, κείμενα αναφοράς, γνωρίζετε την αντίληψή μας. Και να σας πω ότι η δημιουργία της υπηρεσίας αυτής, καθώς και της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων, θα μας επιτρέψουν να εντατικοποιήσουμε την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία όσον αφορά την διαχείριση κρίσεων και σχεδιασμού από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Κιάν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που θα σας πω σήμερα βασίζονται σε κάποια έκθεση που πέρσι ε, δημοσίευσε το, το, το Ίδρυμά μας την πρώτα δέκα χρόνια της CSTP ε, και ε, ΚΕΠΑ και, και έχουμε 23 τέτοιες ε, επιχειρήσεις της περσινής χρονιάς μπορούσαμε να καλύψουμε και κατόπιν ε, αντίστοιχα κάποια γενικά συμπεράσματα. Για να σας πω τι προκύπτει αυτή την έκθεση πάντως. Για καθένα από αυτά τα συμπεράσματα είχαμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι το έχουμε πάρα πολύ καλά, αλλά πάρα πολλές από αυτές μας τις ε, επιχειρήσεις ήταν ε, με μικρής ε, σχετικά κλίμακα, να δούμε το τι έχει οργανώσει η Ένωση τον ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια. Επίσης κάτι άλλο που θα πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι εννοούμε με αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο καθένας έχει και άλλη αντίληψη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κανείς να επειδή άλλο είναι τελειολιστική, σφαιρική, άλλο ολοκληρωμένη προσέγγιση και όλα αυτά ε, ανάλογα με την οπτική γωνία σημαίνουν άλλα πράγματα. Και είπαμε για τον Άτο γιατί ακριβώς υπήρχε πρόβλημα να μπορέσουν να καταλήξουν σε, σε, σε μια τέτοια ολοκληρωμένη ε, αντίληψη. Ε, βέβαια και για το Αφγανιστάν είχε καταφανεί ακριβώ το ότι μπορεί να υπάρχει πολύ γνώμη. Τώρα όσον αφορά την ε, ε, ΚΕΠΑ, έχουμε την Βοσνία, ε, Κόσοβο και εκεί προσπαθήσαμε να έχουμε αυτή την ολοκληρωμένη σφαιρική προσέγγιση. Πάντως νομίζω ότι περισσότερες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποίησαν αυτή την σφαιρική προσέγγιση. Γενικά όμως είναι αποδεικτό ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τα πάμε καλά γιατί έχουν πάρα πολλούς πόρους και θα πρέπει να τα πάμε ακόμα καλύτερα ή στο μέλλον. Όπως είπε ο προλαλής σας. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το ότι έχουμε κάνει τόσες επιχειρήσεις αλλά πάρα πολλές από αυτές έγιναν με κάποιο τρόπο πάρα πολύ καινοτόμο σε σχέση με την παραδοσιακή αντίληψη των πραγμάτων και να σας πω ότι, ότι συμπεράσματα έχουμε εντλήσει, τι μαθήματα ε, μας δόθηκαν. Ε, τέσσερα τέτοια θέματα ε, έχουν σχέση με αυτή την σφαιρική αντίληψη και προσέγγιση. Ό,τι Didier σας, ήδη σας είπε, πρέπει να καταλαβαίνει κανείς τον πολιτικό σκοπό κάθε φορά που κανένα θα πρέπει να βρει μια κρίση να, ή να παρέμβει σε μια τέτοια κρίση. Θα πρέπει κανείς να είναι ξεκάθαρο για το σε σχέση με το τι πολιτικού στόχους έχει. Είναι σαφές ότι Όσο πιο μεγάλη σύγκληση από τέτοιων απόψεων υπάρχει, τόσο πιο πιθανότητε επιτυχία. Είναι αντίθετα. Και αντίστροφα, εάν δεν είναι ξεκάθαρο το τι, τι επιδιώκουν τα κρατημέλη, αν δεν έχουν συσπρωθεί όλοι πίσω από αυτή την θέση, τότε οι επιδόσει θα τείνουν να είναι χειρότερε. Αυτό ίσχυσε και ήταν αποστολή στο Αφγανιστάν. Μια που δεν υπήρχε η πολιτική υποστήριξη, τα ήταν αντίστοιχα για την Παλαιστίνη ε, και εκεί πέρα υπήρχε πρόβλημα. Αν θέλει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική, αν θέλει να ασχίζει περισσότερη επίδραση σε σχέση με όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ε, δαπανά, θα πρέπει να καταβάλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια όσον αφορά τον προβληματισμό του πολιτικά. Τι θέλει, τι πρεσβεύει για όλε αυτέ τι επιχειρήσει η Ένωση. Επομένω, μια συγκεκριμένη πρόταση που εμεί διατυπώνουμε στην έκθεσή μα ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερε κινήσει όσον αφορά ε, την αξιολόγηση, τη μελέτη των καταστάσεων πριν την επανέμβαση. Γιατί θα πρέπει ομένω κάποιο να εξασφαλίσει ότι η εντολή να είναι χρήσιμη και ότι οι πόροι αντιστοιχούν με τι επιτόπου ανάγκε. Αυτό δε είναι ιδιαίτερο ε, σημαντικό για να κανείς έχει ε, επιχείρηση και με πόρους ε, πολιτικούς και στρατιωτικούς. Ιδίως σε την περίπτωση επομένως. Τι χρειάζεται να πετύχει κανείς, πότε χρειάζεται να πετύχει επομένως και θα πρέπει όλα αυτά να συνδέονται με τους πολιτικούς στόχους που θέλει για να συναπατήσει μια τέτοια κατάσταση. The second general lesson and this is maybe a more difficult subject at this particular time, is coherent. Υπό τη σημερινή συγκυρία ακριβώ θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου είδου συνέπεια μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι θα έχουμε. Θα ανοίξουν πύλε του παραδείσου τέλο πάντων με την καινούργια την ε, συνθήκη τη ε, Λισαβόνα. Ε, εδώ, εδώ θα γίνουν όλα αυτά. Είδατε και τα είπαμε και στου Αμερικανού την περσμένη εβδομάδα. Προσπαθούμε να του εξηγήσουμε τι γίνεται. Να, με όλο το σεβασμό προς το, σκόντα. Αντί να έχουμε διαθεσή μα δύο σκόντα θα έχουμε μία σεντέ. να την παραπιβελτίωση του, του υλικού. Ιδίω για τι επιχειρήσει και αυτό. Και θα πρέπει να μην το ξεχνούμε ότι δεν θα πρέπει να εξαρτώμεθα μόνο από τα θεσμικά όργανα για να μα λύνουν τα προβλήματα, θα πρέπει να βελτιώνουμε το πόσο σφαιρική είναι η προσέγγιση. Όμω, όπως και τα μηχανήματα. Ο εξοπλισμό το ίδιο και θεσμικά όργανα. Και άρα και από εκεί μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μα. το πλαίσιο τη διαχείριση. Όπω ξέρετε, είναι εμβαλωματική η προσέγγιση, όπω είπε και ο Ντικία. Και πολλές φορές ήταν τελείως ε, στο γόνατο η προετοιμασία, αλλά και εκ των ενόντων η αντιμετώπιση. Με μια μεριά είχαμε τα κρατημένη που δρούσαν στο πλαίσιο και πάλι, και από την άλλη την Κομισιόν. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν ούτε του μένω ούτε του δε. Αλλά έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανεί να κάτσει και να συνδυάσει όλο τον κόσμο που μπλέκεται. Βλέπετε επομένω ότι τώρα έχουμε ευκαιρία το ώστε όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει επομένω ε, με, με, την, με CMPD όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε την διάθεσή μας. στρατηγείο επιχειρησιακό, στρατηγικό. Δεν είναι ξεκάθαρο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χώρα. Ε, αν θα είναι πολιτικές αρχές, μαζί και στρατηγικές ή χωριστά. Αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μεταξύ του επιτελείου του επιχειρησιακού και της ιστορικής ηγεσία δεν είναι πάντοτε οι καλύτερες. Δεν υπήρχαν πάντοτε οι καλύτερες σχέσεις για κάθε περίπτωση τώρα. Όσον αφορά τους πόρους, ξέρετε ότι για κάθε πολιτική χρειάζεται όσο για να έχει κανείς περισσότερους πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς. Αυτό είναι κοινό μυστικό. Όμως υπό τη σημερινή οικονομική συγκύρια και την κρίση δεν είναι θέμα να βρει κανείς νέους πόρους. Είναι το πώς θα χρησιμοποιήσει τα όσα έχει διάθεσή του και μάλιστα καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό ισχύει και για την αναπτυξιακή βοήθεια. αλλά λάβουμε υπόψη και τι έχει ξοδέψει στο παρελθόν η Κομισιόν. Για κάτσουμε και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Όλοι λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανα στρατιώτη συγκεκριμένο ποσό αναπτυξιακή βοήθεια. Α, στο Αφγανιστάν. Πολύ καλό παράδειγμα. Πολύ περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια σε Βοσνία παρά σε Αφγανιστάν και ίσω γι' αυτό και τα πήγαμε τόσο καλά στο Αφγανιστάν όπω στη Βοσνία. Πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τους πόρους να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι υπάρχοντε πόροι. Και για τον στρατιωτικό εξοπλισμό, ξέρετε, εκεί τα πήγαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά κάποιες περικοπές, ας πούμε όσον αφορά τους κληρωτούς που κατεβήκαν κατά 80%. Όμως η εξοικονόμηση αξιοποιήθηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. 1,9 εκατομμύρια έχουμε διαθεσή μας. Αλλά μπορούμε να αναπτύξουμε και να υποστηρίξουμε το 5% 100.000. Ε, αυτό δεν είναι αρκετό. και το 70% των δυνάμεων ξηρά στην Ευρώπη. Επομένω, οι διεθνεί επιχειρήσει είναι άχρηστοι. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και επίση θα κάνουμε και με το πολιτικό προσωπικό. Εκεί βέβαια οι δυνατότητε είναι πολύ πιο σημαντικέ Γιατί στο στρατικό μέτωπο εκεί πέρα τα πάμε καλά όσον αφορά την, ε, το, το, το, το υλικό, τον εξοπλισμό, αλλά για να βρούμε πολιτικό προσωπικό είναι πολύ πιο δύσκολο. Βέβαια, ξέρετε, αυτό δεν είναι πρώτη φορά που εμφανίζεται. Δεν μπορώ να πω ότι το κλίμα τώρα βοηθάει στο να έχουν κάποιο είδου μόνιμη δομή συνεργασία. Απλώς δεν λέω να τάξουμε νέους στόχους, αλλά να πετύχουμε αυτούς που έχουμε ήδη ορίσει. Και μετά βλέπουμε. Τελική μου πρόταση. Πάρα πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις τη σημερινή ημέρα. Εταιρικέ σχέσει. Βεβαίω μαζί με τον ΝΑΤΟ για Κόσοβο, για Αφγανιστάν και με τον ΟΗΕ σχεδόν για όλες τις επιχειρήσεις τους περισσότερου και από τον Όμως η αλήθεια είναι ότι πάντοτε δεν ήταν τέλειες οι σχέσεις μας, αλλά εάν θέλουμε, ας πούμε στις μεσεντές που σχέσεις μας τι κάνουμε εμείς σερβι μόνοι μας, καλύτερα να συνεργαστούμε με τους άλλους εμπλεκομένου. Από πάση απόψεις. Λόγω του Αφγανιστάν προέκυψε το θέμα των σχέσεων Ένωσης ΝΑΤΟ. Επίσης, συνεργασίες με τρίτες χώρες για τις ε, επιχείρησει. της ΚΕΠΑ. Η Τουρκία είναι ένα κλασικό παράδειγμα τη συνεργασία με τρίτη χώρα με Ρώσους, ε, Κινέζους, Αμερικανούς ε, στην Σομαλία. Δεν θα πρέπει να τα λέμε όλα μαύρα. Υπάρχει κάποια ακτίνα ελπίδα. Υπάρχουν και κάποια άλλοι σημαντικοί εμπλεκόμενοι. Γιατί ασχολούμαστε με τις δυνατότητε που έχουμε, με την σφαιρική προσέγγιση. Αλλά στην Ιούλεξ του Κόσοβο συμμετέχουν οι Αμερικανοί. Συμμετέχουν και στην επιχείρηση για το κράτος δικαίου και στο Αφγανιστάν. Όμως, τον μπαλάκι στο δικό μας γήπεδο να πάνε πράγματα καλύτερα. Βέβαια, η σφαιρική προσέγγιση δεν είναι πιο δόκιμη σε όλες τις επιχειρήσεις. Όμως, έχουμε κάνει κάποια τέτοια, κάποιες διαπιστώσεις. Η ΔΕ Ένωση προσπαθεί αυτά όλα να εφαρμόσει και στην Βοσνία και αλλού. Υπάρχει ολόκληρη περιπτωσιολογία σε σχέση με την τωρινή αποστολή, την Αταλάντη. Και το πιο βασικά είναι ότι αυτή τη αρχή έγινε μια μεγάλη προσπάθεια κανεί να μπορέσει να συνομιλήσει, να έχει επαφή με την Κομισιόν για τι σχετικέ δαπάνε τη Σομαλία. Είπαμε και πριν για Κορέα, Κίνα, Ρώσους. και έπρεπε να αρχίσουμε και αρχίσαμε την Ουγγάντα. Οπότε είχαμε τέτοιου είδους ε, σφαιρική προσέγγιση με την επιχείρηση Αταλάντη. Εδώ θα πάρω τελεία πρόεδρε, και θα τα πούμε αργότερα. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πολύ περιεκτική παρουσίαση. Ο κύριος Γκόαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Υποεπιτροπή για την πρόσκληση που μου να ομιλήσω σήμερα εδώ. Όπως αναφέρατε, εγώ ήρθα εδώ από τη Νέα Υόρκη, γιατί βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη και συνήθως παρακολουθώ τα Ηνωμένα Έθνη, τη διεξαγωγή ειρηνευτικών επιχειρήσεων εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά επίσης η προσοχή μου στρέφεται και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσω να σας αναφέρω κάποια διδάγματα από την εμπειρία μας στα Ηνωμένα Έθνη να την περάσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν σχέση με τη διεξογή ενεργητικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να πούμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά την συχνότητα αυτών των επιχειρήσεων και το μέγεθο των επιχειρήσεων, πολύ περισσότερα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν 10.000 πολιτικό προσωπικό σε όλο τον κόσμο και 10.000 προσωπικό στην αστυνομία. Και θα ήθελα να αναφέρω του αριθμού, ε, αλλά θα ήθελα να πω ότι και η ποιότητά του είναι υψηλή. Βεβαίω τα Ηνωμένα Έθνη κάνουν και διαπράττουν και πολλά σφάλματα ε, δυσχέρειες, τις στο Σουδάν, αλλά κάνουν και πολλά σωστά πράγματα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η αποστολή στην ΑΕΤ παρά τις ε, δυσκολίες και την ε, καταστροφή της ε, ηγεσία στην ΑΕΤ, παρόλα αυτά σημείωσε μια επιτυχία. Και θα πρέπει να τους ε, περνέσουμε για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Θα πρέπει να είμαστε ταπεινόφρονες, θα πρέπει βεβαίως να ξέρουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη. Σήμερα διεξάγει 23-24 επιχειρήσεις ε, στον κόσμο και θα πρέπει να πούμε ότι 15 από αυτές τις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, δεν θα πρέπει μόνο να έχουμε εταιρικέ σχέσει με, με του άλλου οργανισμού, αλλά θα πρέπει να βρούμε κάποια διδάγματα από του άλλου οργανισμού. Και νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα από τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη είναι κάτι το οποίο επεσήμαναν και ο Ντάνιελ και ο Ντιντιέ. Και αυτό είναι το ότι δεν έχει νόημα να μιλούμε για πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, δεν έχει νόημα να μιλούμε για την οικοδόμηση της ειρήνης ή για μια σφαιρική προσέγγιση. Ε, παρά με, με την προπόθεση ότι έχουμε μια πολιτική στρατηγική. Θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους και θα πρέπει να έχουμε κατά νου ποια είναι η τελική κατάσταση στην οποία επιθυμούμε να δεύσει μια χώρα. Εάν δεν το κάνουμε, οι αστυνομικέ δυνάμει είναι άχρηστε, τα στρατεύματα είναι άχρηστα και οι πολίτε είναι άχρηστοι. Γιατί όλα αυτά, όλοι αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο τα εργαλεία εξυπηρέτηση μια τέτοια πολιτική στρατηγική. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, μια επιχείρηση που ήταν εξαιρετικά προβληματική και για τα Ηνωμένα Έθνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή είναι η κοινή αποστολή της ΕΟΦΟΡ στο Τσάντ. Ε, κοινή αποστολή, όπω είπα, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Ηνωμένων Εθνών στο Τσάντ. Έγινε μια προσπάθεια, όπω είπε ο Διντιέ, για να δημιουργηθεί μια σφαιρική προσέγγιση στο Τσάντ, τουλάχιστον εκ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι προσπάθειε αυτέ δεν μπόρεσαν να σημειώσουν στρατηγική πολιτική επιτυχία. Οι δυνάμεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αποτελεσματικές από τακτική άποψη, οι στρατιώτες έσωσαν κάποιες ε, ζωές κλπ. Παρ' όλα αυτά, υπήρξε πολύ φτωχός ε, συντονισμός μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Εθνών. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν σημείωσαν καμία επιτυχία στο Τσάντ όσον αφορά την ανάπτυξη ε, του πολιτικού στρατιωτικού προσωπικού και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να φύγει μετά από ένα χρόνο, κάτι που δεν ήταν έτοιμο να κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη. Υπήρξαν πάρα πολλέ εντάσει μεταξύ των δύο πλευρών και υπήρξαν εντάσει μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και τη χώρα που ήταν υπέρ αυτή τη επιχείρηση περισσότερο από όλε τι άλλε χώρε, που ήταν η Γαλλία. Και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Η Γαλλία είχε κάποιου πολιτικού στόχου στο Τσάντ που δεν συμμερίζονταν όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα Ηνωμένα Έθνη. Και ενώ υπήρξε βραχυπρόθεσμα μια ανθρωπιστική επιτυχία, η κοινή ανθρωπιστική αποστολή των ΗΕ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Τσάντ παρέμεινε κατακαιρματισμένη και δεν έκανε πολλά, πολλά πράγματα για να βελτιώσει την ε, αξιοθρύνητη πολιτική κατάσταση στο Τσάντ ή να συμφέρει στη βελτίωση τη πολιτική ε, κατάσταση. Όπω είπε ο Ντάνιελ, δεν υπήρξε πάντοτε σφαιρική προσέγγιση. Ωστόσο, ορισμένε φορέ είχαμε και ορισμένε φορέ είχαν κάποιε επιχειρήσει που δεν είχαν ξεκάθαρου πολιτικού στόχου. Και το αποτέλεσμα ήταν διασπάθηση χρημάτων ε, και, προσ... Ε, και κατασπατάληση των προσπαθειών. Τι άλλο μπορούμε να διδαχθούμε εξετάζοντα αυτέ τι εμπειρίε ε, με ξένο ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πιο σημαντικό, ε, το πιο σημαντικό πράγμα σε κάθε ειρηνευτική αποστολή είναι το ζήτημα της ηγεσία. Γιατί μπορεί να έχετε όλους τους θεσμούς, τον προγραμματισμό και τις δομές, αλλά χωρίς καμία αποτελεσματική πολιτική ηγεσία δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική μια τέτοια αποστολή. Το σύστημα των μένων εθνών τη πολιτική ηγεσία είναι διαφορετικό από αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εκείνοι αναπτύσσουν στρατιωτικέ ε, ή αστυνομικέ δυνάμει σε μια χώρα, αποστέλουν και έναν ειδικό εκπρόσωπο τη Γενική Γραμματεία που είναι επιφορτισμένο με όλε τι δραστηριότητε των ΗΕ στην ελόγω χώρα. Τι πολιτικέ δραστηριότητε, τι δραστηριότητε στρατιωτική ανάπτυξη και τι αστυνομικέ δραστηριότητε. Είναι ένα είδο ε, είναι ένα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ε, γενική ηγεσία. Και με τον τρόπο αυτό ε, υπάρχει και μία εποπτεία πάνω στον εξοπλισμό και τα μέσα τα οποία βρίσκονται στη διάθεσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολουθεί αυτή τη στρατηγική. Υπάρχουν ειδικοί εκπρόσωποι που δίνουν κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, αλλά δεν έχουν τον έλεγχο των αστυνομικών και στρατιωτικών ε, δυνάμεων. Και υπάρχουν κάποια χάσματα και λήψει. Ε, ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει μια διαφορετική ηγεσία των δυνάμεων που αποστέλλονται από τα Ηνωμένα Έθνη και αυτών που αποστέλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που οδηγεί εν τέλει σε κατακαιρματισμό και σε μια αύξηση τη σύγχυση. Για παράδειγμα, στη Βοσνία η U4 στο παρελθόν έκανε κάποιες επιχειρήσεις πάταξης του εγκλήματος ε, χωρίς να ενημερώσει τις αντικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, καταρχήν, ε, και νομίζω ότι θα έπρεπε να αποσταλεί ένα μήνυμα καλύτερου συντονισμού. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο βήμα, γιατί εάν δεν υπάρχει μια ηγεσία, όσο και καλά προγραμματισμένη είναι η στρατηγική, τελικά θα εκφυλιστεί και θα κατακαιρματιστεί. Και ε, γίνεται πολλή συζήτηση αυτή τη στιγμή εν σχέση με το ρόλο των ειδικών, των είπα των εκπροσώπων μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύσουμε το ρόλο μα και να μην του υπονομεύουμε. Αυτό είναι σημαντικό για τη χάραξη τη πολιτική τη Βρυξέλλε και για τη χάραξη τη πολιτική στο επίπεδο του Συμβουλίου. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε πολλέ επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάρα πολύ καλέ στρατηγικέ στα χαρτιά, αλλά τελικά ε, λόγω τη πολιτική παρέμβαση εκ μέρου των χωρών ε, μελών σημαίνεται αποτυχία. Για παράδειγμα, ε, στο Κόσοβο όπου πήγα δύο φορές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και αξιωματούχοι από άλλους ε, οργανισμούς ε, παραπονέθηκαν ότι ορισμένοι ήταν υπέρ της ανεξαρτησίας του Κωσόβου και άλλοι που ήταν κατά της ανεξαρτησίας του Κωσόβου και τελικά χάθηκε ε, πάρα πολύ χρόνος για προσπάθειες παρέμβασης στο, επίπεδο, ε, στο ίδιο το Κωσυβοπαίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ τελικά έπρεπε να ληφθεί δράση, αλλά όλοι ήταν αντιστακτικοί γιατί εάν έκαναν, έπαιρναν, την πλευρά, έπαιρναν τη μία πλευρά θα προσέβαλαν τους Βρετανούς, αν έπαιρναν το μέρος της άλλης πλευράς θα προσέβαλαν τους Ισπανούς. Η ULEX ε, είχε και θετικά αποτελέσματα, αλλά τελικά η πολιτική παρέμβαση υπήρξε ιδιαίτερος επιζήμια. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι προσεκτικά τους ώστε να μην υπάρχει αυτή η υπονόμευση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας των χωρών μελών. Ο Τιτιέ είπε πολύ σωστά ότι δεν έχει νόημα να σταθεί μια στρατηγική για τις αστυνομικέ δυνάμεις ε, χωρίς ε, να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουν. Ορισμένες φορές οι στρατιώτες αστυνομικοί αλλά και οι πολίτες ε, γίνονται αντιδραστικοί. Τελικά θέλουν δηλαδή να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα, να εφαρμόζονται παροχημένα ή μάλλον τα προηγούμενα μοντέλα, μοντέλα που αποδείχθηκαν επιτυχημένα, να τα επαναλάβουν και την επόμενη φορά. Και πολλέ φορέ γίνεται η προσπάθεια μα Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδημιουργηθούν στρατηγικέ και πολιτικέ που λειτουργήσαν αρκετά καλά στη Βοσνία, επί παραδείγματι, να επαναληφθούν. Αλλά αν εφαρμοστεί η στρατηγική που εφαρμόστηκε στη Βοσνία, εφαρμοστεί στο Αφγανιστάν, ε, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα γιατί η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική. Ή αν θέλετε ε, να επαναλάβατε τη στρατηγική του Κοσοπεδίου στο Κονγκό και πάλι ε, τα αποτελέσματα δεν θα είναι καλά γιατί οι συνθήκε είναι διαφορετικέ. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξει επανάληψη στρατηγικής ε, άλθεια στο Κόσοβο. Ε, η επόμενη γενιά των Ευρωπαϊκών Αποστολών ε, ίσως θα πάει στην Ιεμένη, σε χώρες της Βόρειας Αφρικής, όπου έχει ενισχυθεί η παρουσία της Αλκάιντα. Θα αποστείλουμε στρατιωτικό προσωπικό οι πολίτες εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος από τρομοκρατικές υποθέσεις ε, επιθέσεις. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στα παλιά και παροχημένα μοντέλα. Ε, νομίζω να έχουμε μια δυνατότητα νέου προγραμματισμού, του να προσαρμοστούμε καλύτερα στα νέα περιβάλλοντα. Θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους ε, άντλησης διδαγμάτων. Τα Ηνωμένα Έθνη έχει μία μονάδα 50 ανθρώπων που προσπαθούν να αντλήσουν κάποια διδάγματα από τι ρέχου επιχειρήσει, κάτι το οποίο δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μετά την καταστροφή τη Βοσνία στο 1990, τα Ευρωπαϊκά Έθνη άσκησαν μεγάλη αυτοκριτική και ήταν ειλικρινή όσον αφορά τα ίδια του τα σφάλματα. Ενώ εμεί ε, στι ε, Βρυξέλλε δεν είμαστε ιδιαίτερω ε, κριτικοί στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη το 2000 εξάδωσαν μία έκθεση ε, η οποία ε, προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια μιας αναπροσαρμογής των στρατηγικών της. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί για τις μελλοντικές ειρηνευτικές αποστολές προσπαθώντας να επεξεργαστεί την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά να δει τι γίνεται και σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει υποστεί πάρα πολλές ε, μεταβολές και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα έχετε πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, ακριβώς από αυτού θα εργαστούμε εδώ, γιατί η επόμενη μας έκθεση που θα γίνει από, εδώ, από την Επιτροπή μας δηλαδή θα αφορά ακριβώς την ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πολιτικοστρατηγική συνεργασία ε, και σίγουρα ε, όσοι θα συντάξουν έκθεση θα εξετάσουν όλες αυτές τις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα. Τελευταίος ο μιλητής ο κ. Μέλινγκ. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ είμαι σε μια πολύ καλή, βρίσκομαι σε πολύ καλή θέση. Οι προηγούμενοι ομιλητέ απλώ σα τα έπανα όλα. Εγώ απλώ μπορώ να κλείσω, να συνοψίσω και αν δεν αρκεί αυτό, να πω απλά πω υπάρχει μια μελέτη που έχουμε κάνει, ένα ενημερωτικό έγγραφο και αν χρειάζεται περισσότερε λεπτομέρειε, βρίσκονται όλε εκεί. Ε, αλλά οι συνάδελφοι ούτω ή άλλω ε, ήταν πολύ περίεκτικοι. Αυτό το ενημερωτικό έγγραφο που φτιάξαμε ε, έπρεπε να περιλαμβάνει μια ειδική προοπτική όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων από τις Ένωσες γιατί δηλαδή ε, και αν χρειάζεται να έχει τέτοιες δυνατότητες η Ένωση, μέσα στο πλαίσιο των πρόσφατων διδαγμάτων που έχουμε αποκομίσει, καθώς και το μεταβαλλόμενο στρατηγικό περιβάλλον, δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ε, ιδέες, από θεσμικούς τριγμούς και ε, τριβές καθώς και από πρόβλημα όσον αφορά την ε, παροχή πόρων. Υπάρχει δηλαδή χώρος για βελτίωση επιτόπου. Η συνθήκη της Λισαβόνας που τώρα έχει αρχίσει να ισχύει και είναι βέβαια επαρκής ε, αλλά όχι μάλλον απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή αλλαγή και καινοτομία. Και αυτό γιατί οι, τα θεσμικά όργανα δεν φτιάχνουν την πολιτική. Και βέβαια εκτός αυτού όλοι ανέμεναν ε, ότι περιμένουν ότι διάφορες κρίσεις αμφισβητούν τις δυνατότητες της Ένωσης πλέον για την οικοδόμηση ειρήνης. Θα, ορισμένοι συνάδελφοι λένε ναι, χρειάζεται πολιτική για την οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας και πρέπει εμείς να το σκεφτούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ένωσης, ποια μέσα έχει στη διάθεσή της για να το επιτύχει όλα αυτά εν γέννη δηλαδή πώς μπορεί, μια στρατηγική, πώς, πώς μπορεί να είναι μια στρατηγική για την οικοδόμηση της ειρήνης από πλευρά της Ένωσης. Δεν υπάρχει μια απλή στρατηγική που να μπορούμε να πούμε ναι αυτό θα κάνουμε και σίγουρα θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Και ακόμη περισσότερο όταν υπάρχουν πολλές διαφορετικές πολιτικές και όχι μία. Και γι' αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα μια, μια συζήτηση όσον αφορά το ενδιαφέρον και την αξία των προτεραιότητων που θέλουμε να επιτύχουμε. Δηλαδή μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση δικά τη συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο αντιστρόφω ανάλογα. Βασικά λοιπόν έχουμε την οικοδόμηση ειρήνης, δηλαδή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την οικοδόμηση ειρήνης και δεύτερον η δομή και ε, η οργάνωση, δηλαδή ποιος κάνει τι και γιατί. Από την πλευρά τη θεσμική εμείς ε, έχουμε μεγάλη γραφειοκρατία. Αυτό σημαίνει από τη μια πλευρά θα πρέπει να συνδέσουμε τα βραχυπρόθεσμα με τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, οι αστυνομικές αποστολές, ε, ε, σχεδιασμός, εφαρμογή, όλα αυτά θα πρέπει να συνδεθούν γιατί, πρέπει... γιατί φαίνεται να υπάρχει μεγάλο κενό ανάμεσα στα δύο. Για τους πόρους, ε, τονίσαμε ότι ίσως θα ήταν καλό να συγκεντρώσουμε τους πόρους και έτσι να περιορίσουμε την γραφειοκρατία, γιατί η γραφειοκρατία δεν, δεν της αρέσει γενικά η συγκέντρωση των πόρων. Ωστόσο, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις όπου η γραφειοκρατία έχει βρει πολύ παραγωγικές και εφάνταστες λύσεις. Θα πρέπει βεβαίω να λάβουμε υπόψη και την ανθρωπιστική πτυχή. Τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει την στρατηγική οικοδόμηση ειρήνη. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία που έχει για να μπορέσει να μεταβάλει το σύστημα Καταρχήν θα πρέπει να παρουσιάσει μια εικόνα για το ποια θα πρέπει να είναι μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και να, να, να εξασφαλίσει πως τα αποτελέσματα αυτά θα μπορέσουν να ελοκληρωθούν στη διαδικασία οικοδόμησης των νέων δομών, τόσο εντός των Βρυξελών, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο του 2012-2013. Και επίσης ε, οι απαραίτητες υπηρεσίες της Κομισιόν να είναι ολοκληρωμένες ή τουλάχιστον υπόλογες στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων να υπάρχει δηλαδή μια ευρύτερη ε, προσέγγιση όσον αφορά την οικοδόμηση ειρήνης και επίσης να γίνεται καλύτερη χρήση των εμπειριών της Κομισιόν στην εφαρμογή. Ο ύποπτος εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλες τις απαραίτητα, όλα τα απαραίτητα μέσα για να εξασφαλίσει την συνοχή των πολιτικών ε, ε, μοντέλων και στόχων και θα ήθελα να δώσω έμφαση στο τι είπε ο για, τον, εκπρόσωπο, για τους ειδικού μάλλον εκπροσώπους της Ένωσης. Ορισμένοι θέλουν να τους, εξεφ, να ε, περιβάλλοντά τους με, μεγάλ, με, με γραφειοκρατία. Αυτό που μπορούμε να μάθουμε από τον ΟΗΕ ε, ωστόσο, εγώ πιστεύω είναι ότι ο ειδικό εκπρόσωπο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο δεδομένου του κύρου του επιτόπου. Είναι πάντα πολύ δύσκολο, εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε φορά, αλλά υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Και για τις γραμμές του προπολογισμού Εν γέννη νομίζω πως είναι απαραίτητο μακροπρόθεσμα να είμαστε υπέρ της εξέτασης της συγκέντρωση των κονδυλίων. Το Κοινοβούλιο να εκτιμά τον προπολογισμό και την δαπάνη των ε, κονδυλίων με βάση τις προτεραι... στρατηγικές προτεραιότητες. Το να έχει κάνει στρατηγική σημαίνει να έχει και κάποιο κανόνα για να μπορεί να κρίνει. Να μπορεί, μπορείς εκ των προτέρων ακριβώς να κρίνεις τι θα κάνουν τα θεσμικά όργανα και οι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί στη διεκπαιρέωση όλων αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για τις τέσσερις αυτές εισηγήσεις που πιστεύω ότι θέτει τη συζήτηση στα θεμέλια. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους για την πρώτη φάση της συζήτησης, να κάνω μια ερώτηση και ίσως και ένα σχόλιο που κατά κάποιο τρόπο είναι και ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση αφορά συγκεκριμένα τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν τα μέσα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των παλαιότερων συζητήσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με την έκθεση που κάναμε για την PSDC, Κάποιε φορέ επικρατεί η καχυποψία, είτε πολιτικέ επιφυλάξει και ιδεολογικέ επιφυλάξει, αλλά και οργανωτικέ επιφυλάξει όσον αφορά αυτό το συνδυασμό των πολιτικό-στρατιωτικών. Επικρατεί δηλαδή ο φόβο ορισμένε φορέ ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε ένα είδο στρατικοποίηση των δομών. Για πολιτικούς λόγους ορισμένες χώρε είναι ουδέτερες, για ιδεολογικούς λόγους άλλες φορές άλλες είναι... Ε, πολλοί βουλευτές λοιπόν έχουν υπογραμμίσει αυτό το κίνδυνο τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβανόμεθα, αντιλαμβάνονται ορισμένοι ως κίνδυνο. Ήταν λοιπόν ένα ερώτημα, τι, τι θα συμβεί και πώς θα διοργανωθούν όλα αυτά πιο συγκεκριμένα στις δομές που έχουν φτιαχτεί και η συνεργασία πώς γίνεται, ποιο είναι το ιστορικό των ανθρώπων που είναι εκεί και επίσης όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό. Η στρατιωτική είναι εξοπλισμένοι για όλα αυτά. Μήπω είναι περισσότερο εξοπλισμένοι από τους πολιτικούς που μπορεί να εργάζονται στι ίδιε δομές. Τι συμβαίνει, σε Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και θα επανέλθω στο δεύτερο μου παρατήρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ ώρα για αυτή την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι είναι κάπως δύσκολο να καταλάβω αυτή την προβληματική γιατί για το δικό μας φορέα είναι πάρα πολύ εύκολο. Προτείνουμε στο Συμβούλιο κάποιους στόχους ανάλογα με τους πολιτικούς στόχους της Ένωσης, οπότε το ερώτημα είναι να δούμε με τι μέσα θα πετύχουμε πιο πρόσφατα το στόχο μας. Και λέμε ότι συνήθως αυτά είναι τα στρατιωτικά μέσα, σε κάποιες φορές, άλλες φορές όμως, χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν πόροι πολιτικοί. Οπότε θα, η κάθε φορά, ο κάθε φορά προγραμματισμός εξαρτάται από κάποια ανάλυση που έχει γίνει ήδη. Τώρα, όσον αφορά το ΣΕΜ5 και τη συγκρότησή του, διάβασα και εγώ τι τις εφημερίδες και με απασχόλησε το θέμα. Όσον αφορά αυτούς τους 25 υπαλλήλους, όχι 23 συγγνώμη, αυτούς που απασχολούμε στην υπηρεσία μας. Έχουμε 10 εξ αυτών οι οποίοι έχουν ένα background ε, το οποίο, προέρχονται από στρατιωτικό κλάδο ή από το διπλωματικό κλάδο και ε, έχουν ήδη απασχοληθεί σε κάποια ερευνητικά κέντρα 10-10 από αυτούς τους υπαλλήλους οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους ε, παρελθόν και έχουμε άλλους 7 στρατιωτικούς οι οποίοι υπηρετούν σε αυτή μου την ε, μονάδα και άλλους έξι που έχουν ε, παρελθόν ε, νομικό ή έχουν υπηρετήσει σε αρχές, αστυνομική. Και αυτοί λοιπόν οι προγραμματιστές ευκολότερα μπορούν να λειτουργήσουν. Άλλωστε, περισσότεροι από αυτούς τους προγραμματιστές είναι, στην αγορά από στρατιωτικό παρελθόν παρά πολιτικό. Με προϋπηρεσία δηλαδή στις στρατιωτικές αρχές. Οπότε, όταν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης από αυτή την εξωτερική υπηρεσία, τότε θα κινηθούμε και προς ε, αυτές τις δύο ε, κατευθύνσεις. Είπαμε 10 διπλωμάτες ε, και 6, 7 ε, στρατηγοί και 6 νομικοί αστυνομικοί πρόεδρος. Αυτό που εγώ ήθελα να σας πω αφορούσε αυτό που τονίσατε ότι πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσουν αυτές οι επιχειρήσεις και να πετύχουν αυτές οι ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρο πολιτικό στόχο τον οποίο να σπάζονται όλα τα κρατημέλη τα οποία θα συμμετάσχουν. Αλλά η δυσκολία είναι, παρά το ότι συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε, είναι το πώς θα γίνει διαχείριση της κρίσης. Εκεί που προκύπτει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική συνένεση. Για να μην πάμε σε χειρότερη αποτυχία. Γιατί υπάρχουν κάποιε επιχειρήσει που αποφασίζονται υπό το κράτο του κατεπήγοντος. Άρα, πώς θα κρυθεί αυτό. Α πούμε, υπάρχει ηθική επιταγή να πανέβει κανεί. Α πούμε, στα Βαλκάνια δεκαετία του 90. Ήταν, ήταν κάτι το κατεπήγον. Συμφωνούν όλοι ούτω ώστε να είναι δυνατόν στρατηγικά να θεωρηθεί ότι υπάρχει συνένεση. Ιδάλλως κανείς να μην ε, επέμβει. Γιατί την άλλη μεριά μπορεί κανένας να μην έχει τη συνένεση, να, να παρέμβει, αλλά έτσι να μπορέσει να περιορίσει τις ε, κακές συνέπειες. Οπότε όταν δεν υπάρχει το κατεπήγον, μπορεί κανείς να έχει το περιθώριο να βρει την τη συνένεση όπως το κρυσφοπαίδιο. Είχαμε 22 συν 5. 22 θέλαν την ανεξαρτησία, την αναγνώριζαν και άλλοι 5 όχι. Παρ' όλα αυτά, οι και οι 27 συμφώνησαν όσον αφορά την αποστολή. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε συνένεση με ενιαίο όραμα όσον αφορά την αποστολή. Άρα, πώς θα συνδεθεί το ένα θέμα με το άλλο, η συνένεση με την ε, ανάγκη της επέμβασης, όπως ας πούμε έχει γίνει στην περίπτωση της Γεωργίας. Δεν υπήρχε ούτε τότε σύμφωνη μεταξύ των 27. Πώς θα απαντούσετε εσείς για αυτή την αντίφαση. Από μια μεριά δηλαδή ο χρόνος που πιέζει και από την άλλη μεριά το πόσο επίγον είναι κανείς να επέμβει σε σχέση με το ότι χρειάζεται συνένεση. Κύριε Λούνατσεκ, έχετε πρώτη το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και εσάς για, την, ε, για τις παρεμβάσεις σας. Ε, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ντανζάν. Δηλαδή η ανάγκη της χάραξης μιας ξεκάθαρης πολιτικής στρατηγικής και ενός ξεκάθαρου πολιτικού στόχου. Κάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει σε πολλούς τομείς, δεν υπάρχει με αυτή την καθαρότητα. Εγώ η ίδια είμαι συγγήτρια για το κοσυφοπαίδιο και το αναφέρατε κι εσείς ο ίδιος. Και εδώ είναι ένα από τα σημαντικά προβλήματα, ότι σε πολλές από τις αποστολές και το, στο τσάτ συνέβη κάτι παρόμοιο. Υπήρξε το πρόβλημα ότι σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρξε ξεκάθαρος πολιτικός στόχος. Και έτσι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόζονται σε πολιτικο-στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε να είναι. Ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορείτε να απαντήσετε αυτό το θέμα, δηλαδή πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η δική μας πολιτική σε σχέση με αυτή την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ξεκάθαρη δήλωση εκ μέρου σας είναι σημαντική, γιατί είναι κάτι που εγώ ίδια το γνωρίζω, αλλά είναι χρήσιμο να ακούμε και από εσά πως η έλλειψη ξεκάθαρων πολιτικών στόχων, και αυτό το βλέπουμε συγκεκριμένα στο Κωσυφοπαίδιο, τελικά οδηγεί στην κατασπατάληση των πολλών κονδυλίων, ε, των πόρων, του εξοπλισμού κλπ. Ε, και δεν ε, οδηγεί σε μια εφαρμογή 100%. Το συγκεκριμένο μου ερώτημα πηγαίνει στην κατεύθυνση ενός θέματος το οποίο αναφέρθηκε εδώ το εξή. Οι περισσότερες από τις αποστολές είναι πολιτικού χαρακτήρα. Για μένα, όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης ε, της Λισαβόνας, ε, εδώ προβλέπεται ένα σημαντικό στοιχείο, η πρόληψη. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε να κάνουμε για να ενισχύσουμε αυτή την ε, πολιτική πτυχή, την μη στρατιωτική πτυχή. Δηλαδή να μην ε, περιμένουμε να δεχθούμε στην κλιμάκωση των συγκρούσεων, αλλά να δρούμε στο επίπεδο της πρόληψης. Είπατε στον προγραμματισμό δεν έχουμε επαρκές προσωπικό και όταν υπάρχει προσωπικό είναι περισσότερο στρατιωτικό. Τι πρέπει να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη μη στρατιωτική πτυχή, την πολιτική πτυχή και να έχουμε μια δυνατότητα μη στρατιωτικού προγραμματισμού. Ε, κύριε Λενουάρ, μας εξηγήσατε τι γίνεται με το δικό σας επιτελείο, την αναλογία πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού. Τι κάνετε από τη δική σας πλευρά για να ενισχύσετε το, μη το μη στρατιωτικό σκέλος. Λέτε ότι γίνονται εδώ λίγο στα πράγματα, αλλά πού εντοπίζετε εξής ακριβώς τα ελλείμματα και τις δυνατότητες παρέμβασης. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα. Ε, βλέπουμε ότι η τάση πηγαίνει προς την ενίσχυση των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αλλά στις χώρες μέλη, στις περισσότερες χώρες μέλη, ε, υπάρχει, δεν υπάρχει η διάθεση να αποστέλλονται ε, στρατιώτες, στρατιωτικές δυνάμεις, ε, γιατί είναι υψηλό το κόστος, γιατί θέλουν να αφήσουν τις χώρες αυτές να βγουν μόνες τους από, από τα προβλήματά τους. Πού λοιπόν ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει παρόλα αυτά η ανάγκη αποστολή στρατιωτικού ε, προσωπικού στρατιωτικών δυνάμεων και πού βλέπετε ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό εφόσον υπάρχει όπως είπαμε αυτή η τάση μείωσης εδώ μείωση του στρατιωτικού σκέλους. Στην Ευρώπη έχουμε διατυπώσει από κοινού το αίτημα να υπάρξει ένα τμήμα οικοδόμησης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ε, και αυτή τη στιγμή η κυρία Άστον και το Συμβούλιο ε, λένε ότι ίσως δεν χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο, ε, να υπάρξει ένα φιδελές τμήμα. Αλλά θα πρέπει όλα τα τμήματα να ασχολούνται με αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό είναι το ίδιο όπως γίνεται με την ενίσχυση της θέσης των γυναικών, το gender mainstreaming. Ε, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει ένα ανεξάρτητο τμήμα το οποίο να ασχολείται ειδικά με αυτό το θέμα. Το ίδιο ισχύει και για την οικοδόμηση της ειρήνης. Θα πρέπει να υπάρξει μια αυτοτελής ε, δομή για την οικοδόμηση της ειρήνης που να μεριμνά να συμπεριλαμβάνεται η πτυχή αυτή σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα και τι κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Λούζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντόνατσεκ τελικά με επικάλυψε σε πολλά σημεία. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Λενουάρ. Μας περιγράψατε πώς είναι τα διάφορα, διάφορες μονάδες, διάφορα τμήματα, διάφορες τομείς. Κατά την άποψή μου δεν θα υπάρξει πλέον αυτοτελής πολιτικός ε, σχεδιασμός. Τι λέτε για την κριτική του Αλέν Τετρού από την ομάδα για τη διεθνή κρίση ε, που λέει ότι η διαχείριση των κρίσεων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει μία στρατιωτική κατεύθυνση. Λέει ότι κινούμεθα προς ένα μέλλον όπου οι στρατιωτικοί υπερογνώμονες τελικά αναλαμβάνουν το σχεδιασμό πολιτικών αποστολών, πολιτικών επιχειρήσεων. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο έγινε σαφές στην τελευταία παρουσίαση, όπου είπατε ότι υπάρχουν περισσότεροι από το, στο στρατιωτικό τομέα απασχολούνται με το ζήτημα του προγραμματισμού. Εγώ έχω σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες και ασχολούμαι με, την, ε, με ζητήματα υγείας, σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και εδώ δεν υπήρχε ούτε ένα στρατιωτικό. Πώ είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο πολλοί στρατιωτικοί που να ασχολούνται με θέματα προγραμματισμού, Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, τομεί καθαρά πολιτικού χαρακτήρα. Εάν από τη δική σα πλευρά παρουσιάζονται έτσι τα πράγματα, λέγεται δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι που ασχολούνται με τον προγραμματισμό από το στρατιωτικό τομέα και ακούμε όλο και περισσότερο διατυπώσει όπω επιχειρήσει, αυτή για μένα δεν είναι μια θετική ένδειξη για την ενίσχυση των πολιτικών αποστολών στο μέλλον. Αντίθετα, οι αναλύσεις μάλλον θα γίνονται μελλοντικά κάτω από ένα στατικό πρίσμα. Η κυρία Λούνατσεκ αναφέρθηκε για παράδειγμα στο ζήτημα του φύλου τις θέσεις των γυναικών. Και διαρωτώ με πώς οι στρατιωτικοί μπορούν να διαπιστώσουν ακριβώς τις υφιστάμενες δομές στην ΑΕΤ, ότι εκεί υπάρχουν πολύ ματριαρχικές ε, δομές και οι γυναίκες έχουν έναν ενισχυμένο ρόλο στην κοινωνία των πολιτών. Πώς είναι δυνατόν οι στρατιωτικοί να αξιοποιήσουν αυτές τις δομές, για παράδειγμα, για να φροντίσουν για μια βιώσιμη και αποτελεσματική αυτοοργάνωση της κοινωνίας της ΑΕΤ. Ε, κυρία Γκόν, ε, ε, στη μελέτη σας προτείνετε κάποιους στόχους όσον αφορά την αύξηση του στρατιωτικού δυναμικού των χωρών ε, μελών. Γιατί λέτε ότι οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτυχάνουν αυτούς τους στόχους θα πρέπει, στις χώρες αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται ορισμένε κυρώσεις. Θα μπορούσατε να μου πείτε τι είδου κυρώσεις φαντάζεστε εδώ. Και το τελευταίο ερώτημα έχει ως εξής. Προτείνετε τα battle groups να μετατραπούν σε στρατιωτικές δυνάμεις. Θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια ενίσχυση της ε, πολιτικής ε, διάστασης που να αντικαταστήσει αυτά τα battle groups ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ βλέπω εδώ με μεγάλο ενδιαφέρον το σημερινό έγγραφο από το Συμβούλιο και έχω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Ποιο στυλ επικρατεί εδώ σε αυτές τις πρώτες φάσεις, αλλά και όχι στις πρώτες σελίδες, αλλά όχι μόνο σε αυτό εδώ το έγγραφο, αλλά γενικά στα όλα τα έγγραφα που προκύπτουν το Συμβούλιο για το τι θα πρέπει να γίνει και το Ελπίζω πως θα έρθει κάποια στιγμή. όπου θα διαβάζουμε τέτοια πράγματα, όπου θα λέει ότι το Συμβούλιο καλωσορίζει το γεγονός ότι δεν χρειάζεται πλέον να επαναλάβει προηγούμενα σε θεωρίες και αιτήματα. Και μετά βλέπω ας πούμε τι λέει για την κατάσταση στη Γεωργία. Το Συμβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του κτλ. κτλ. Μα ποια εργαλεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το Συμβούλιο για να πετύχει τους στόχους. Το να επαναλαμβάνει είναι κούφια λόγια. Ορισμένοι λένε πως είναι καλύτερο να μιλάνε παρά να σιωπούν. Αλλά όταν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Υπάρχει επίσης μια θέση που λέει διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανά μέσα στα διοικητικά όρια και ότι αυτό είναι κλειδί για την οικοδόμηση της, οικοδομ... της εμπιστοσύνης. Πολύ ωραία και καλά όλα αυτά. Αλλά πώς θα επιτευχθεί αυτή η πρόοδος για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης Πώς προτίθεται να λάβει μέτρα που να προωθήσουν την πρόοδο στην εξέβρεση του κλειδιού για αυτή την κατάσταση, χωρίς καν να λέει το όνομα της ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να υπάρξει καμία πρόοδος. αν δεν υπάρχει πρόοδος, το να λέμε απλώς ε, λόγια δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση στο Κάφκασο. Σε σχέση με τις αγώνες που προβλέπεται να γίνουν εκεί, τι ε, αθλητικές εκδηλώσει που θα γίνουν εκεί. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Äh, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση σε σχέση με τόσα υπόθηκαν από διάφορες πλευρές, δηλαδή ότι θα πρέπει στην αρχή κάθε δράσης να υπάρξει, να προηγηθεί ένα, μια ξεκάθαρη στοχοθεσία. Αυτό μου θυμίζει τα όσα είπε ο Γερμανός ο φιλόσοφος και λογοτέχνης ο Εφραίμ Λέσιγκ ε, από την εποχή του διαφωτισμού με τίτλο για την ε, βαθμιαία ανάπτυξη των ιδεών κατά την ομιλία. Νομίζω ότι το αίτημα αυτό, το οποίο διατυπώθηκε εδώ, ε, κατά κάποιο τρόπο είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα, ενώ ε, στην πραγματικότητα πρόκειται για την ε, βαθμία ανάπτυξη των σκοπών κατά την εφαρμογή. Θεωρώ λοιπόν ότι όσον αφορά το ζητούμενο θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να υπάρξει ένα ξεκάθαρος στόχος, κάτι το οποίο θα μας βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία αναφέρατε κι εσείς. Νομίζω εγώ ότι το ζητούμενο θα ήταν πώς ε, στο πλαίσιο μιας τέτοιας αποστολής η θεματοποίηση και η διαφάνεια των αντιφάσεων μπορεί να εξασφαλιστεί. Δηλαδή, εάν πράγματι υπάρξουν κάποιες δυσκολίες στον ορισμό των στόχων ή στην εφαρμογή των στόχων, ε, κάτι που ε, απειλεί να παρεμποδίσει την επιτυχία μια δράση, πώ μπορεί να φροντίσει ούτω ώστε οι συγκρούσει αυτέ να γίνουν αντικείμενο διαχείριση, αποτελεσματική διαχείριση και να εξασφαλιστεί η διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτή είναι σημαντική. Ε, αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Λενουάρ καταρχήν. Αναφέρατε μια στατιστική όσον αφορά την ε, κατανομή των ε, προσώπων που συνεργάζονται μαζί σας και έχουν διάφορες ε, ειδικότητε, προέρχονται από διάφορους τομείς και θα με ενδιαφέρει να μας πείτε κατά πόσο υπάρχει εδώ μια ιεραρχία, δηλαδή πώς κατανέμονται αυτοί οι νομικοί, οι διπλωμάτες ε, σε σχέση με τους ε, στρατιωτικούς. Αν θέλουμε να τα δούμε εδώ ιεραρχικά, να κάνουμε μια ιεράρχηση. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνατε θα σχηματίσαμε μια κάπως διαφορετική εικόνα. Και μια παράκληση. Είναι καλό εάν ε, κάποιος γνωστοποιεί το γνώσο ότι ε, μας χρησιμοποιεί κάποιου αριθμού για κρίσιμα θέματα. Αλλά όταν χρησιμοποιούνται κάποιοι αριθμοί, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όλοι οι αριθμοί, όχι μόνο ορισμένοι αριθμοί που τελικά συμβάλλουν στο να δώσουν μια εξορισμένη εικόνα. Και επίσης να διαφοροποιήσετε το διπλωματικό και στρατηγικό προφίλ. Τι εννοείται ε, ε, στρατηγικό προφίλ. Είναι σαν συνάρτηση με κάποιες στρατιωτικές ειδικότητες. Και ένα τελευταίο ερώτημα σε σχέση με την ε, πλειονότητα των δράσεων που ήταν ε, πολιτικού χαρακτήρα, μη στρατηγικού χαρακτήρα. Μπορώ να φανταστώ ότι τέτοιου δράσει στο επίπεδο του προγραμματισμού μπορούν να επωφεληθούν από αυτή την πολιτικο-στρατηγική συνεργασία. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αξιολόγηση τυχών κινδύνων που μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα η στρατηγικοί από τους πολιτικούς εμπειρογνώμενους. Αυτό μπορώ να το φανταστώ απολύτως. Αλλά ταυτόχρονα φαντάζομαι ότι σε κάποιο σημείο, για παράδειγμα, ανακύπτει μια δυσκολία για καθαρά πολιτικές δράσεις και υπόθηκε εδώ ότι μελλοντικά θα υπάρξουν περισσότερες τέτοιες πολιτικές δράσεις. Όταν εδώ ε, στρατηγικοί εμπειρογνώμονες τελικά είναι αρμόδιοι, έχουν τελευταία λέξη και για πολιτικές δράσεις. Πώς μπορούμε δηλαδή από τη μία να αξιοποιήσουμε το νόχα, την τεχνονοσία των στρατηγικών, από την άλλη να παρεμποδίσουμε στρατηγική με την δική τους ε, δική συγκεκριμένη νοοτροπία ε, και ματιά να επικυριαρχήσουν και να στρέψουν τα πράγματα στη δική τους κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που ενδείκνεται για καθαρά πολιτικές δράσεις. merci. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, το ζήτημα αυτό αναφέρθηκε εδώ πολύ πλατιά από πολλούς ομιλητές. Ποιος θέλει να απαντήσει, ίσως οτι Διντιέ Λενουάρο στον οποίο απευθύνθηκαν πολλά ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις ετέθηκαν για το πώς ε, θα συνδυάσουμε τον επίγοντα χαρακτήρα και την ανάγκη συγκέντρωση συνένεση. Υπάρχουν δύο είδη συνεργασία. Πρώτον, εκεί που υπάρχει απόλυτη συνένεση των 27 για όλε τι 27 χώρε και πραγματική βούληση να προχωρήσουμε. Αυτό θα ήταν το ιδανικό υπάρχει όμως και η άλλη που όπου υπάρχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται σε, για κάποια συγκεκριμένη κατάσταση και που ενδιαφέρονται για το ότι αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό δεν χρειάζεται να, αποτελ... να αποκλειστεί. Τα δυο μου πρότυπα αυτά μπορούν να είναι συμπληρωματικά. Βέβαια πάντοτε να ζητούμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και την πιο εις βάθος συνένεση, τόσο το καλύτερο θα ήταν αυτό, αλλά εάν τα κράτη που θέλουν να αντισταθούν, που θέλουν να αντισταθούν πρέπει να τους αφήσουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί αυτό αποτελεί ε, τμήμα της ευελιξίας μιας διεθνούς οργάνωσης. Για το θέμα της πρόληψης των κρίσεων, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Με ρωτήσατε Ποιες ήταν οι υπόψεις μας για το θέμα αυτό. Φυσικά είναι ένας στόχος που αποτελεί τμήμα των θεμελιωδών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Να επιμένει όσο γίνεται περισσότερο στην πρόληψη των συγκρούσεων. Δεν υπάρχει εδώ καμιά αμφιβολία. Εκεί όπου μπορεί να υπάρξουν αποκλήσεις θεμητές όσον αφορά τις εκτιμήσεις είναι με το ποιο τρόπο θα διασφαλίσουμε την λειτουργία και την παρακολούθηση αυτών των θεμάτων πρόληψης των κρίσεων. Υπάρχει δυνατότητα να θεσπιστεί μια διάκριση ανάμεσα στην πρόληψη συγκρούσεων, την διαχείριση των κρίσεων και την επιβολή της ειρήνης. Υπάρχει επίσης και η λογική που λέει ότι η πρόληψη των συγκρούσεων, αν αποτύχει, θα πρέπει αμέσως να περάσει κάτι πιο στεναρό, και άρα υπάρχει και η νομιμότητα να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι ο ρόλος της πρόληψης των συγκρούσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πρόληψη. Η... αποστολές εκπαίδευσης αστυνομικών ή στρατιωτικών που κάνουμε είναι πρόληψη, πρόληψη των κρίσεων κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει λοιπόν πιστεύω αμφισημία όσον αφορά την ε, προσήλωσή μας στην διαχείριση των κρίσεων. Αυτά μπορώ να πω για την ώρα. Για τώρα το ερώτημά σας, το τι κάνω για να έχω περισσότερους πολιτικούς εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να είμαι ειλικρινής, δεν κάνω τίποτα, γιατί χρειαζόμαστε δημοσιονομικές θέσεις, θέσεις στον προπολογισμό και το ξέρετε πολύ καλά καλύτερα από μένα ότι αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο μιας συμφωνίας δημοσιονομικής. Ένας θεωρητικός πίνακας προσωπικού έχει βέβαια φτιαχτεί και προβλέπονται διάφορες θέσεις για πολιτικούς και θα τις καλύψουμε μόλις θα έχουμε στην διάθεσή μας τα απαραίτητα κονδύλια. με ρωτήσατε πώς αντεδρώ για ένα άρθρο, νομίζω είπατε, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαταλείπει τις δραστηριότητες διαχείρισης κρίσης λόγω του ε, της λειτουργίας του CMDP. Πιστεύω πως αυτό είναι μια κρίση, αλλά στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι δραστηριότητες της μονάδας μου από τότε που δημιουργήθηκε Είμαστε στην στρατηγική έκθεση για το Αφγανιστάν, για το Ιράκ. Εργαζόμαστε για την Γουινέα Μπισάου και για το Κονγκό. Ε, δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εγκαταλείπει φυσικά την πολιτική διαχείριση κρίσεων. Κάτι τέτοιο είναι παράξενο. Η πραγματικότητα επιτόπου θα μας οδηγήσει στο τι θα κάνουμε. και αν χρειαστεί να διαχειριστούμε κρίσεις θα τις διαχειριστούμε. Προσπαθώ να αποφύγω τη λέξη operation, επιχείρηση, και χρησιμοποιώ τη λέξη mission, αποστολή. Σίγουρα δεν θέλω να δώσω καμία στρατηγική γεύση σε οποιαδήποτε πολιτική ε, επιχείρηση. Για τις στρατηγικές και πολιτικές πτυχές θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν κατάλαβα ακριβώς ποια είναι η ερώτησή σας. Ο ΙΕ αναπτύσσει πολύ περισσότερους ε, στρατικούς από ότι αστυνομικούς. Δηλαδή δεν είναι η προέλευση του ανθρώπου που ορίζει τις ικανότητές του. Ε, εξαρτάται αυτό από τον τρόπο τον οποίο έχει εκπαιδευτεί το, στα διαδρομία του και ούτω καθεξής αλλά υπάρχουν και γίνονται κάποιες ε, ειδικέ καταρτήσεις πριν την ανάπτυξη όλων αυτών των αποστολών. Και εξάλλου οι στρατιωτικοί που χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιούνται γιατί έχουν συνηθίσει να συνεργάζονται με τους πολιτικούς και με τους πολίτες. Οι στρατιωτικοί συνήθω εκπαιδεύονται στο να αντιμετωπίζουν και την κατάσταση των ε, αμάχων εκεί όπου βρίσκονται. Τώρα, για το τι χρειάζεται να γίνει στην γεωργία και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δικές μας ενέργειες εκεί. Ε, φυσικά και δεν πρόκειται να σας πω ότι 100% πετυχαίνουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί εγώ περνάω 12-13 ώρες την ημέρα προσπαθώντας να λύσω όλες αυτές τις δυσκολίες και ξέρω πως υπάρχουν προβλήματα και όλοι γνωρίζουμε το περίφημο την περίφημη ρίση της ε, Αμερικανικής κυβέρνησης που λέει ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα το οποίο να αντιστέκεται στην πραγματικότητα της ζωής. Είμαι ο τελευταίος που θα σας πω ότι όλα τέλεια τα καταφέρνουμε. θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Γεωργία μπορούμε ίσως να εξετάσουμε ε, διαφορετικές λύσεις να μου πούμε τι, θα είχε γίνει αν δεν είχε υπάρξει ευρωπαϊκή ε, παρέμβαση. Θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνω το μήνυμά σας και γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Για το δικό σας ερώτημα για την κατανομή εντός της δικής μου ομάδας. Έχω τέσσερις επικεφαλής θρηματάρχες. Δύο είναι στρατιωτικής προέλευσης και δύο πολιτικής. για το θέμα του ότι οι στρατιωτικοί έχουν τον τελευταίο λόγο στο σχεδιασμό. Αυτό, δεν, λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη αν έδωσα τέτοια εντύπωση. Προετοιμάζουμε έγγραφα για το Συμβούλιο. Οι υπουργοί κάνουν τι επιλογές τους και εκείνοι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Και δεν υπάρχει στρατιωτική παρέμβαση στην πορεία. Κανένας από τους δημοτάρχες δεν είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις νομίζω. Εμείς κάνουμε σχεδιασμό. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη χρήση των πόρων που έχουμε, των πολιτικών πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Φυσικά και θα βελτιωθούμε, βελτιωνόμαστε ε, και θα βελτιώσουμε τους πολιτικούς μας πόρους γιατί συμφωνώ μαζί σας πως ε, εδώ έχουμε πρόβλημα και Όλα αυτά αποτελούν ε, τμήμα του σχεδιασμού του εξωτερικής υπηρεσίας. Δεν θέλω να μπω τώρα στις λεπτομέρειες, αλλά δεν υπάρχει καμία όρεξη από πλευρά του στρατιωτικού τομέα να αναλάβει και το πολιτικό. Αυτά έχω να σας πω για την Ευχαριστώ. Έχετε εσείς να πείτε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σύντομα δύο λόγια για το κατά πόσο μπορεί να προγραμματίσει αυτή την ταχεία επέμβαση. Η αντίδραση που εσεί το είπατε, Πρόεδρε, γιατί όλοι καταλαβαίνουν το πόσο δύσκολο είναι τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν για μια κοινή θέση. Για οτιδήποτε. Ιδίω αν υπάρχει μια τέτοια κρίση, από τι οποίε πρέπει να επιληφθεί κανεί. Όμω, όπω έχουν τα πράγματα με αυτή τη θεσμική συζήτηση που γενικά γίνεται για το τι θα γίνει με τα τέλη αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τουλάχιστον να μπορέσουμε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερα, καλύτερα πλαίσια, καλύτερα θεσμικά ε, εργαλεία για να λάβουν οι απόψει, γιατί άμα λάβουν την απόφαση τα κρατημέλη να μπορέσουν να δράσουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ε, ακριβώς το να υπάρχει το CMPD. Βέβαια η Βαρονία, Άστον και όλη η εξωτερική υπηρεσία βέβαια θα βοηθήσουν, αλλά αποσχεληθεί η απόφαση να υπάρχει το πλαίσιο, να υπάρχουν δυνατότητε, να υπάρχουν θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν για να υπάρξει δράση. Δεύτερον, όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων, νομίζω ότι πάρα πολύ σωστό είναι το ότι ετέθη το θέμα του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η καλύτερη πρόληψη παρά ε, η θεραπεία και ε, πρόσφατα έχουν περίπου 5% μέχρι το, έως το 2013 συγκεκριμένα το 2008 που έχουν δαπανηθεί για αυτήν την πρόληψη των κρίσεων. Όμως μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα και δεν μιλώ ε, για ανθρωπιστικές δαπάνες, μιλώ για αναπτυξιακή πολιτική. Ανάλογα επομένως όπως είπαμε με τις ε, με, τις, με τους στόχους που έχουμε, να δούμε επομένω πώς μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων της πολιτικής της ε, αναπτυξιακής. Ε, θα πρέπει όμως αυτό να οπωσδήποτε να ξανασυζητηθεί τώρα όσον αφορά αυτούς τους 100.000, παμε 70.000 70-80.000 ε, από αυτούς που έχουμε στη διάθεσή μας ε, τους αναπτύσσουμε, επομένως δεν έχουμε και πάρα πολλούς που να περισσεύουν για αλλού, Αφγανιστάν, Βοσνία, Κόσοβο και δεν μπορώ να απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Στρατηγικά πώς να σου απαντήσω και ο κόσμος μας αλλάζει συνέχεια. Οπότε βλέπουμε ότι οι ΙΠΑ όλα και περισσότερο προσέχουν την ασφάλεια στην Ασία και όχι μόνο στην ε, Μέση Ανατολή. Για να κοιτάξουμε και εμείς την γειτονιά μας και δεν είναι μόνο Κάφκασο, Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια, μιλώ και για της Σαχάρας, μιλώ και για Ινδικό Ωκεανό και στη Γαλλία είχαν φτιάξει έναν ε, χάρτη ε, και, και φτάνανε όσον αφορά λέγανε το ενδιαφέρον κομμάτι ε, μέχρι και πέρα από τη Ρωσία και μέχρι την Νότιο την Αφρική, νοτιούς της Σαχάρας. Εμάς αυτό είναι πάρα πολύ πάρα πολύ ρεαλιστικό. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω σενάρια ιδιαίτερα για Κάφκασο κλπ. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι ρεαλιστικά, αν τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο. Με δύο λόγια όσον αφορά την πολιτική. Τι λέγανε Beatles. All you need is love. Το μόνο που χρειάζεται κανεί είναι αγάπη. Όχι, το μόνο που χρειάζεται κανεί είναι πολιτική θα λέγαμε. Για τη δική μα περίπτωση. Ε, Αναφέρατε και την περίπτωση της ε, Γεωργίας, γιατί όλοι ξέραν τότε ότι ήταν πάρα πολύ πιθανό να ξεσπάσει πόλεμος και μας το λέγανε αυτό οι του ΟΗΕ από το 2005-2006. Ε, ένα σωρό ε, δημοσιεύματα υπήρχαν στην Tribune, τα έλεγε ο Χόλμπρουκ και άλλοι και άλλοι όσον αφορά το πόσο πιθανό. Δεν ξέρω φυσικά πότε θα ξεσπάσει Ούτε ξέραμε πόσο γρήγορα θα κέρδιζαν οι Ρώσοι, αλλά ξέραμε ότι είναι κάτι πολύ πιθανό να ξεσπάσει ο πόλεμο. Και γνωρίζαμε φυσικά ε, το πού θα κατέληγε αυτό ο πόλεμο. Ε, και αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα του πώς κανείς μπορεί να προλάβει τις εξελίξεις. Να μπορέσει εκ των προτέρων να αποφασίσει τι θα κάνει όταν ε, συμβεί κάτι. Οπότε και στο Τσάδ ισχύει το ίδιο. Ότι η διεθνή παρουσία εκεί θα ωφελούσε τον Τριστέμπη. αυτό θα βγει κερδισμένο. Τα ξέραμε αυτά. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αναφορές αλλά δεν έχουν το χρόνο αυτοί οι κορυφαίοι να τα διαβάσουν. Και για το Κόσοβο ξέραμε ότι θα γίνει εκεί η έκρηξη, ξέραμε ότι υπήρχε διαφθορά όμως πήρε δύο χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσω τι θα κάνω, εγώ μπορούσα να σα το, πω από το 2001. Άρα είναι θέμα πολιτικών προγνωστικών. Άλλο πολιτικά προγνωστικά και άλλο σχεδιασμός επιχειρησιακός. Αλλά εδώ είναι η ουσία της πρόληψης των κρίσεων. Αν κανείς μπορεί να έχει προγραμματισμό και πληροφορίες, μπορεί και να προλάβει για τις κρίσεις. Δύο λόγια τώρα σε σχέση με το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια ε, προ... πρωτοβουλία πολιτικής αντίδρασης Ευρώπης. Έχουμε αυτούς που θα θέλανε να πάνε στην εμπολεμιζόνη δεν τους αφήνουν. Ναι, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει νόμος και είναι φτύνο το ποτό. Προσοχή, επομένω, μην πάνε εκεί πέρα λάθο άνθρωποι με αυτού του είδου την πρωτοβουλία. Αλλά θα μπορούσαμε όμω να συγκροτήσουμε ένα σώμα με κάποιου ε, οι οποίοι να, είναι, να ξέρουν την, την επιμελητία, να ξέρουν ε, όλα τα σχετικά. Ε, λίγες εκατοντάδες. Αλλά αυτή θα είναι η χμή του δόρατος για οποιοδήποτε είδους ε, πολιτική, ε, πολιτικό φορέα, πολιτική δύναμη. Και κατόπιν με αρχή και βάση αυτούς προχωράμε. Σαν τον Jedi στο Star Wars. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο, επικεφαλή. The final point, um, civilian military balance. Τώρα όσον αφορά την, το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ στρατιωτικών, στρατιωτικού προσωπικού και πολιτικού όσο δημοκρατικό και να είναι στρατός, θα πρέπει να υπάρχει, ε, να υπάρχει κάποια, κάποια αναλογία πολιτικού προσωπικού στι Βρυξέλλες και επί τόπου. Γι' αυτό και εγώ και συναδελφοί τονίζουμε το πόσο χρήσιμο είναι να υπάρχει συμμετοχή του ευρωπαϊκού υψηλού εκπροσώπου. Όπως ο Πίτερ Φάστο Κόσοβο μπόρεσε να κάνει περισσότερο με 200 ε, ε, αστυνομικούς παρά όλη η ένοπλη δύναμη έκανε. Πρόεδρος. Δίνει το λόγο στον ε, κύριο Μέλινγκ. Όλοι μιλούν για τη διαφορά, το κοινό, αυτό που χωρίζουν από πολιτικούς, πολιτικό προσωπικό από στρατιωτικό, όμως κανείς δεν λέει τη διαφορά μεταξύ του πολιτικού προσωπικού. και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μας αυτή η διαφορά ότι ακόμα και όταν υπάρχει ένας στατιώτης υπάρχει αυτός ο διχασμός, η αντιπαράθεση. Υπάρχουν αντιμαχόμενα συμφόρα. Συμφέροντα κάποιοι έχουν κάποιες ιδέες καινούργιες, άλλοι θέλουν να φροντίσουν τη διατήρηση ειρήνης, Τώρα, στρατηγική διαχείριση κρίσεων, πρόληψη. Δεν μπορεί κανείς να κάνει προγνωστικά, μπορεί όμως να δει συμπεράσματα. Και ξέρουμε, ενώ δουλεύουμε σε μια κρίση, μαθαίνουμε κάποια πράγματα, Και κάθε φορά γινόμαστε και καλύτεροι. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει η τέλεια στρατηγική. Είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρίς να υπάρχει κάποια στρατηγική. Είναι δυνατόν να αρχίσει κανείς μια επιχείρηση χωρίς κάτι να έχει προσχεδιάσει. Um, on Για το αν χρειάζονται στρατιωτική. Όχι, δεν αποφασίζουν αυτοί. Οι κυβερνήσεις συμπληρώνουν τους στρατιωτικούς με το πολιτικό προσωπικό. Έχουμε τους προγραμματιστές, έχουμε τους γιατρούς, έχουμε τους μηχανικούς. από τις θεωρητικές σχολές όμως και τους θέλουν αυτούς να βοηθήσουν τους θεωρητικούς. Δεν ξέρουμε, δεν είναι το άριστο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι το θέμα του πόσο ενδιαφέρουσα είναι σαν δουλειά αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψατε μου να σας πω ότι είναι αυτό ακριβώς το θέμα του προγραμματισμού. Μπορεί κανείς να ε, ε, προβλέψει ότι θα υπάρξει μια σύγκρουση στη Γεωργία παραδείγματι και θα πρέπει να προετοιμαστεί. Εγώ θα ήθελα να πω το θέμα είναι, το είναι η πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί και για τον προγραμματισμό. Το 2002 είχα μία θέση στη Γενέβη, στα Ηνωμένα Έθνη, όταν επίκει το πόλεμο του Ιράκ όλοι γνωρίζαμε τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσει ένας προγραμματισμός πριν ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας γιατί θα ασκείται στην περίπτωση αυτή η δρυμία κριτική. Το ίδιο ισχύει και για το Κωσυφοπέδιο. Εγώ συμμετείχα στη διαπραγματεύση για το καθεστώς του Κωσόβου. Όλοι βλέπαμε ότι θα ερχόταν θα έμπαινε αυτό το θέμα της ανεξαρτησίας του Κωσόβου. Αλλά όταν προσπαθεί να κάνει κανείς ε, προγραμματισμό λέγοντας ότι θα πρέπει μία αποστολή των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντικαταστήσει μία αποστολή των Ηνωμένων Εθνών ενώ ας πούμε τα Ηνωμένα Έθνη σε γραφειοκρατικό επίπεδο αμφίστανται, δεν θέλουν να δώσουν τη σκητάλη στην ΕΟΛΕΞ και υπάρχουν ορισμένε χώρες που δεν θέλουν να το κάνουν και είναι μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ανακύπτουν αυτές οι δυσκολίες. Ε, υπάρχει ε, από τη μία το ζήτημα της ε, πολιτικής απόφασης και από την άλλη το ζήτημα του προγραμματισμού, τα οποία ενδεχομένω είναι σε μια σύγκρουση. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πάλι σε σχέση με τις παρατηρήσεις του Richard Γκάουεν εν σχέση με την εποπτεία του μη στρατιωτικού σκένλους. Ε, θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση σε σχέση με το ρόλο αυτού του κοινοβουλίου. Ε, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα είναι ότι εμείς εκ των υστέρων μετά τις αποστολές αυτές ε, προσπαθούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση. Έχουμε για παράδειγμα την ετήσια έκθεση του Προέδρου ε, για την ε, ΚΕΠΑ και εκεί περιλαμβάνονται γνωμοδοτήσεις και αξιολογήσεις για τις διάφορες αποστολές που βρίσκονται από εξέλιξη. Αλλά πώς φαντάζονται εμπειρογνώμονες συνολικά τον, ε, έναν επαρκή ρόλο αυτού του Κοινοβουλίου εν σχέση με την μη στρατιωτική εποπτεία των εν αποστολών. Ευχαριστώ πολύ και η κυρία Λούνατσεκ θέλει να πάρει το λόγο και στη συνέχεια θα σας δώσω το λόγο για να καταλήξετε και θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα μια διευκρινιστική ερώτηση που να διευκρινίσει ακριβώ αυτή τη σχέση μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών. Ε, είπατε, ε, κύριε Κεβάν, ότι οι δαπάνες ε, για αναπτυξιακή βοήθεια έχουν κάποιες επιπτώσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να μεριμνήσουμε για το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, γιατί αυτό έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια και άλλων περιοχών του κόσμου. Έχω την εντύπωση και από τα όσα είπε ο κ. Λενουάρ ότι δεν κάνει διαφορά από το που προέρχεται κανείς αν έχει ένα στρατικό ή μη υπόβαθρο αν θέλετε αλλά νομίζω και θα ήθελα να πω ότι εγώ η ίδια γνώρισα στρατιωτικούς που πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ γιατί έχουν μια ιδιαίτερη ορθολογική προσέγγιση στις καταστάσεις, πολύ περισσότερο από τους πολιτικούς ορισμένες φορές. Αλλά θα πρέπει το να είναι κανείς να έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να χειριστεί ένα όπλο ή δεν έχει αυτή την κατάρτιση, νομίζω ότι αυτό κάνει μια διαφορά. Επίσης, η αναλογία ανδρών και γυναικών. Θα με ενδιαφέρει να μου πείτε εσείς, ε, κύριε Λενουάρ, στο δικό σας τμήμα, πόσοι, πόσα από τα υψηλά στελέχη, από τους υψηλούς αξιωματικούς, είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα όσον αφορά το επίπεδο πρόληψης των συγκρούσεων, θεωρώ ότι είναι κεντρική σημασία να απασχολούνται εδώ πολύ περισσότερες ε, γυναίκες. Και οι γυναίκε ε, εκπροσωπούνται πολύ περισσότερο στους μη στρατιωτικού τομεί. ξέρετε ε, τη δουλειά που έγινε εν σχέση ε, με, τις, ε, με το τι συμβαίνει σε κάποιους τομείς πριν οδηγηθούμε στην στρατιωτική κλιμάκωση. Έχουν μια σχετικές έρευνες όπου λέγεται ότι ε, οι γυναίκες για σε χωριά όπου ξέρουν που είναι αποθηκευμένα τα όπλα τα οποία ενδεχομένω θα χρησιμοποιηθούν. Και όλες αυτές τις πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να μπορέσει κανείς να προλάβει τι συγκρούση ακριβώς πριν οδηγηθούμε στην κλιμάκωση. Γι' αυτό απευθύνω και πάλι την έκκληση να αυξηθεί η αναλογία των γυναικών, ειδικά σε αυτούς τους τομείς. Και επίσης το ποσοστό των ανδρών που δεν έχουν, που δεν είναι καθαρά στρατιωτική, δεν έχουν μια στρατιωτική εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές για να απαντήσουν και μετά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ. Ε, εντάχει θα απαντήσω την ερώτηση σας, ε, κυρία μου. Στο τμήμα μου υπάρχουν ε, τέσσερα, στην μονάδα μου τέσσερα τμήματα υπάρχουν δύο γυναίκες επικεφαλής και δύο άνδρες. Θα έλεγα ότι εγώ είμαι κάπως ε, απομονωμένος στο δικό μου, δική μου μονάδα, γιατί εκεί υπάρχουν τρεις γυναίκες και μόνο εγώ σαν άνδρας. Ο ρόλος των γυναικών είναι σημαντικός όχι μόνο στο επίκεδο της πρόληψης, αλλά και μετά. Χρειαζόμαστε νοσοκόμε κλπ. Ε, για όλα αυτά είμαι απολύτως ε, πεπισμένος για τη συμβολή των γυναικών δηλαδή. Uh, Chairman. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω αυτά που είπε ο Διδιέ όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ στρατηγικού και μη στρατητικού σκέλου. Ε, νομίζω τα πράγματα είναι πολύ απλά. Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι είναι μυστικό το να δούμε πώς η Ουάσιγκτον προετοιμάστηκε για τον πόλεμο στο Ιράκ. Δεν ήταν οι στρατιωτικοί αυτοί που άσκησαν τη μεγαλύτερη πίεση Ξέρετε τι ακριβώς εννοεί όταν λέει το background ε, ορισμένων ανθρώπων. Ε, δεν νομίζω τα πράγματα είναι πολύ απλά ή απλουστευμένα όπως τα παρουσιάζεται. Εγώ πάντοτε είμαι υπέρ μια σφαιρικής ε, προσέγγισης, θεωρώντας ότι θα πρέπει να είμαστε κάπως ευέλικτοι. Um, the, on... Ναι, όσον αφορά το προγραμματισμό, και τους κινδύνους ε, νομίζω ότι είναι ένα εσωτερικό ζήτημα. Όσον αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου, ε, όσον αφορά την εποπτεία του μη στρατιωτικού σκέλους, ντρέπομαι να πω ότι δεν γνωρίζω πολύ καλά τους κανονισμούς του Κοινοβουλίου για να σας δώσω ακριβείς απαντήσεις. Κάτι που ανέφερα στην αρχική μου παρουσίαση ήταν την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές βρίσκεται πίσω από τα Ηνωμένα Έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά με κάποια διδάγματα που θα έπρεπε να είχε αντλήσει, ιστερή δηλαδή. Δεν νομίζω ότι εξετάζει πολύ προσεκτικά τα διδάγματα τα οποία θα μπορούσαν να αντληθούν από την κάθε αποστολή και από τα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δραματίσει ένα πολύ σοβαρό ρόλο στο πλαίσιο ακροάσεων όπως αυτή αποκτώντας τις περισσότερες ε, δυνατές πληροφορίες ε, εν σχέση με τις υποεξέλιξη ε, αποστολές. νομίζω ότι θα πρέπει, όπως σας είπα, να κοιτάξουμε προσεκτικότερα τα, τις εμπειρίες που έχουμε συγκεντρώσει, τα διδάγματα από το Τσάτ, το Κόσοβο κλπ, όπου τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν εξαιρετικά δύσκολα και νομίζω ότι οι λύσεις που δόθηκαν θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει μια υποεπιτροπή και στην Καπούλ και να δείτε τι μπορείτε να μάθετε εκεί, επιτόπου δηλαδή. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, πιστεύω. Ένα θέμα το οποίο δεν απαντήθηκε στο τελευταίο γύρο, κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ένα, μια αυτοτελή δομή για την οικοδόμηση της ειρήνης. Νομίζω ότι συνδέεται με το ζήτημα του Ιράκ το Ζήτημα της ιεραρχίας, συγγνώμη, εν σχέση με την ιεραρχική διάρθρωση κάποιων γραφειοκρατικών δομών ε, και την, επαρκή σύσταση, την σύσταση επαρκών ομάδων. Ε, επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία των πόρων, να μπορούν να δαπανηθούν ε, αποτελεσματικά. Αυτά είναι τα σημαντικά ζητήματα και όχι κατά πόσο θα πρέπει να υπάρξει μια αυτοτελής ε, δομή. Εάν νομίζετε ότι, εάν βεβαίως θεωρείτε ότι πράγματι η οικοδόμηση της ειρήνης συνιστά προτεραιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω ότι ορισμένε φορέ δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί επικεντρώνουμε την προσοχή μα τόσο πολύ σε μια διχοτόμηση μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους. Ε, ε, ε, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια τόσο άκαμπτη λογική. Είπατε ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου η διχοτόμηση μεταξύ ενός μη στρατιωτικού background και ε, διχοτομήσεων μεταξύ, διχογνωμιών ή αποκλήσεων μεταξύ των διαφόρων χωρών ε, είναι πιο καθοριστική. Ε, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε για τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Έχει γίνει εδώ μια σχετική πρόοδος. Έχουν, έχουμε κάνει συζητήσεις για ε, εκθέσεις που έχουν εγκριθεί. Ε, βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν διαφυσβήτητα έχει να σε ένα σημαντικό ρόλο εδώ και στο επίπεδο των διαφόρων ε, δομών που θα συσταθούν στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Γιατί νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε ακόμα σε εμβρική ε, κατάσταση. Είναι θεμελιώδες λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, συμβολές σας δεν μας εμποδίζει τίποτα να επανέλθουμε στα θέματα αυτά στο πλαίσιο του δεύτερου πάνελ, το οποίο θα ξεκινήσουμε αμέσω και το οποίο θα ασχοληθεί περισσότερο με σκέψεις επιχειρησιακού χαρακτήρα όσον αφορά αυτή τη σφαιρική προσέγγιση και την πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Και θα ήθελα να δώσω ίσως το λόγο πρώτα στην κυρία Κρίλ, εάν συμφωνείτε. Monsieur le Président, euh, Κύριε Πρόεδρε, στο όνομα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που μας καλέσατε να συμμετέχουμε σε αυτή την ακρόαση. Θα ήθελα να κάνω μία πρώτη παρατήρηση, αλλά στην πράξη ο... ήδη αναφέρθηκε λέγοντας ότι υπάρχει έλλειψη ορισμών ε, και επίσης σε σχέση με το τι, ε, πόσοι ορισμοί υπάρχουν. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην βασιμότητα και στους κινδύνους ε, για μια, από μια τέτοια συνεργασία ανάμεσα στον πολιτικό και το στρατιωτικό τομέα, γιατί είναι τομείς που τους γνωρίζουμε πολύ καλά στον Ερυθρό Σταυρό. Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία μια τέτοια συνεργασία, θα ήθελα να υπογραμμίσω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Καταρχήν, η χώρα η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση θα πρέπει να επιλέξει ποιε λύσει θεωρεί ότι είναι οι καλύτερε. Η αναζήτηση λοιπόν τη λύση πιστεύουμε πω ε, ε, εξαρτώνται από την ίδια τη χώρα, όπως άλλωστε ορίζει και το διεθνές δίκαιο που ισχύει για τις ε, κρίσεις. Ε, οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνονται για το, προς το συμφέρον των πολιτών. Δεν θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ένοπλες δυνάμεις ή την χώρα από τη στιγμή που αυτές δεν θέλουν να ενεργήσουν, δεν μπορούν δηλαδή οι ε, ανθρωπιστικές δράσεις να αντικαταστήσουν την πολιτική βούληση. Τώρα, επίσης, συντονισμός ε, θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους διάφορους τομείς, πρόθεση καλής διακήρυσης, δικαστικός τομέα. Σα βέβαια, σας θυμίζω κάποια πράγματα που είναι προφανή. Αναγνωρίζουμε πως τέτοιος διάλογος είναι απαραίτητος για να υπάρξει μια τέτοια ε, συνεργασία, αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση όταν χρειάζεται μεγάλη ανάπτυξη ε, μέσων που μόνο οι στρατιωτικοί μπορούν να αναπτύξουν ε, και μέσα σε μικρό διάστημα. Βλέπουμε με τις συνέπειες διαφόρων σεισμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια και αυτά όλα μας θυμίζουν την ανάγκη παρέμβασης στρατιωτικής εκεί βέβαια μια ολοκληρωμένη τέτοια προσέγγιση με πολιτικοστρατική συνεργασία ε, περιέχει κάποιου κινδύνου. Θα ήταν πραγματικά αυταπάτη να πιστεύει κανεί ότι οι χώρε μπορεί να υπακούν ε, προτεραιότητε τρίτων χωρών ή χωρών ε, ή ακόμα και του ΟΗΕ. Αν όλοι οι στόχοι αποτελούν είναι κοινή, τότε η ανθρωπιστική ενέργεια αποτελεί ένα μέσο, ένα εργαλείο στα χέρια του κράτους. Μόνο όταν είναι δηλαδή συντονισμένες οι προσπάθειες και κοινοί στόχοι. Οι όροι ανθρωπιστική βοήθεια πολλές φορές χρησιμοποιούνται και για την ε, χρήση στρατιωτικών δυνάμεων από πλευράς χωρών οι οποίες δεν θέλουν να φανεί πως συμμετέχουν με στρατιωτικές ε, δυνάμεις σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ένοπλες δυνάμεις της ε, ε, αντιπολίτευσης να χρησιμοποιήσουν και να καλύψουν δικές τους δράσεις και πολλές φορές βλέπουν πως υπάρχει ε, συνωμοσία της Δύσης κατά του Ισλάμ. Ε, μεγάλες συνέπειες λοιπόν για τους δικαιούχους της βοήθειας δεν έχουν πια πρόσβαση γιατί ο Ερθρός Σταυρός διατρέχει πολύ μεγάλο κίνδυνο. Πώς μπορούμε λοιπόν να χρησιμεύσει η δική μας εμπειρία ο Ερυθρός Σταυρός έχει δημιουργηθεί το 1863 όπως γνωρίζετε, θέλει να προστατεύει την ζωή και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα πολέμου και να βοηθ... αυτή η εντολή του έχει ανατεθεί από τα κράτη μέσα στο πλαίσιο της Σύμβασης της Γενέβης το 1977 και 2005. Η περιπλοκότητα βέβαια των ενόπλων ε, σειράξεων οδηγεί στο ότι δεν έχει ο Ερυθρός Σταυρός το μονοπόλιο των ανθρωπιστικών δράσεων και πολλές φορές ε, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο προβλέπει δράσεις ε, που μπορούν να τις αναλάβουν τα κράτη-μέλη ε, να τις αναλάβουν οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός. Κάθε φορά πάντως ε, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια ε, προσπάθεια πρέπει να είναι ανθρωπιστική και αμερόληπτη. Θα είναι όμως όλο ένα και πιο αμερόληπτη όταν καθορίζεται αποκλειστικά από τις ανάγκες των θυμάτων. Έχουμε λοιπόν διακυβερνητικές ε, υπηρεσίες ε, του, ε, του ΟΗΕ και γι' αυτό και είναι μεγάλη η ανεξαρτησία μας. Στις περισσότερες χώρες όπου εργαζόμαστε έχουμε πετύχει συμφωνία και επίσης ασυλία αυτής που χαίρουν, αυτή, αυτή την ασυλία στις οποίες χαίρουν γενικά οι διεθνείς διακυβερνητικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει να προσφύγουμε σε, επίσης σε ε, συνοδείες, πράγμα το οποίο ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία μας. Επιπλέον, είμαστε ουδέτεροι από τη δημιουργία μας, ε, απέχοντας από κάθε ε, σύγκρουση ή αντιπαράθεση πολιτική, στρατιωτική, ιδεολογική και δεν ε, μεταβάλλεται δική μας ε, προσπάθεια ε, από καμία επιρροή. Δεν δέχεται καμία επιρροή. Βασιζόμαστε περισσότερο στη δύναμη της πυθούς, προωθούμε τον διμερή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Μέρη. Αυτό σημαίνει μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα διάφορα μέρη που βρίσκονται σε σύγκρουση. <clears throat> Τώρα, έτσι ώστε ο διάλογος να είναι επικοδομητικός, είναι απαραίτητο τα μέρη της σύγκρουσης να συμμετέχουν και να δέχονται την ανθρωπιστική βοήθεια και έπειτα να υπάρχει μια ιεραρχία, μια αλυσίδα ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε τόσο την, τον πληθυσμό όσο και τους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού. Μια, πλεονεκτήματα έχουμε ε, από μια τέτοιου είδους προσέγγιση, ωστόσο δεν είναι πάντοτε εύκολο να πείσουμε τα συγκρόμενα μέρη για την καλή μας πίστη, την ανεξαρτησία μας και την οδετερότητά μας. Κάτι τέτοιο είναι ε, χρονοβόρο, χρειάζεται μεγάλη υπομονή, μια κακή αντίληψη παρεξηγήσεις και σύγχυση με άλλους φορείς γρήγορα καταστρέφουν αυτό το κεφάλαιο εμπιστοσύνης και θέτουν σε κίνδυνο την ανθρωπιστική αποστολή. Το 2003 δεχθήκαμε επιθέσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, στήχησαν τη ζωή τη σε τέσσερι συναδέλφου. και αυτέ οι επιθέσεις φαίνεται πω ήταν η πιθανή σύνδεση του Ερυθρού Σταυρού με ε, τις δράσεις των ξένων ε, δυνάμεων στο ίδιο πλαίσιο. Για να επανέλθουμε στο Αφγανιστάν να πούμε ότι η σύγχυση που προκαλείται από τις διάφορες στρατιωτικές προπαγάνδες αποτελούν, ε, βρίσκονται στην καρδιά τέτοιων σημαντικών ε, ε, περιστατικών. Η διάκριση με τους υπόλοιπους φορείς ε, γίνεται όλο και πιο δύσκολη από τη στιγμή που γίνονται και στρατιωτικές ενέργειες στις ίδιες ε, περιοχές. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους εκεί να ε, καταλάβουν ποιος έκανε κατασκοπικό έργο πριν από την επίθεση. Ε, Επίση, ε, πρέπει διαρκώ να επιβεβαιώνουμε πω οι δράσει μα ε, είναι δεκτέ από όλε τι πλευρέ τη ε, σύγκρουση και φαίνεται πω οι τελευταίε μα προσπάθειε έδωσαν καρπού. Κατά τη διάρκεια του 2009 μπορέσαμε να παίξουμε το ρόλο μα του ενδιάμεσου και του ουδέτερου μάλλον διαμεσολαβητή που οδήγησε σε απελευθέρωση ε, ομήρων λοιπά Το ίδιο και στη Σρι Λάγκα, χάρη στον ε, μόνιμο διάλογο με τους ε, την κυβέρνηση αλλά και τους τίγρης τα Ταμίλ μπορέσαμε να οδηγήσουμε σε απελευθέρωση πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Όλα αυτά χάρη στο διάλογο όπου βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία Πρόσφατα στο Αφγανιστάν, ένας από τους αδέλφους μας ήρθε σε επαφή με έναν πρώην ηγέτη Μουτζαχετίν που ήταν ε, κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1987 και που σήμερα ως φύλαρχο ε, καταπολεμά την κυβέρνηση Σιζαλή. Ε, είπε πως σήμερα, όπως και πριν από 20 χρόνια, επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρό Σταυρό κάνει προσπάθεια για να περιθάλψει τα θύματα. Ωστόσο, μα προειδοποίησε ότι δεν περίμενε ο Ερυθρό Σταυρό να υποστηρίξει τι απόψει του και τι δράσει του, όπω δεν επιθυμούσε να υποστηρίξουν τι θέσει και τι δράσει του εχθρού. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ε, να γνωρίζετε, ε, γνωρίζετε ότι. Θα το έχετε καταλάβει ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκεται κανείς με τέτοιου είδου συμπληρωμένη προσέγγιση ούτω ώστε να υπάρχει κανένα είδου ε, απομάκρυνση από κάθε είδου ενόπλη παρέμβαση, διότι από τότε που είχαμε τη μάχη του Σολφίνου του 1999 δεν σταμάτησαν οι επαφέ του ΣΕΣΕΡ με με κυβερνήσεις και με ε, αντιπολιτεύσεις ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την, την αποστολή μας, να την εξασφαλίσουμε και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των, του προσωπικού μας και γι' αυτό το λόγο ε, είπαμε ότι υπάρχει ο, ο στόχος είναι του να μπορέσουμε να δουλέψουμε με, με κατανόηση και να πριτανεύσει τελικά το διεθνές δίκαιο και ο ανθρωπισμός ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το δόγμα για την, την παιδεία, την εκπαίδευση και όσον αφορά το Αφγανιστάν ε, είχαμε τακτικές επαφές με τις ε, ένοπλες δυνάμεις, τους Αμερικανούς, το ΝΑΤΟ, το ώστε να υπάρχει ασφάλεια και με αυτόν τον διάλογο μπορέσαμε να ε, να, ε, να, να, να, έχουμε κάποια, κάποια καταγραφή κάποιων περιπτώσεων ε, εγκλημάτων όσον αφορά την, ε, την παραβιάση του διεθνούς δικαίου και για δε το Κονγκό ε, επίσης δράσει τον ίδιο τρόπο ώστε να έχουμε έναν διάλογο διαρκή με την Μονίκ και όσον αφορά το πολιτικό προσωπικό ε, γιατί πέσαν 10 χρόνια ακόμα όλα αυτά είναι και καυτή ε, επικαιρότητα και είπαμε ότι πάντοτε η δράση μας ρυθμίζεται από το διεθνές δίκαιο και εγκατακλείδη θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι πάρα πολύ βασικό ότι η πολιτική, η στρατιωτική και οι ανθρωπιστικοί φορείς οι οποίοι ε, συμμετέχουν στην ίδια επιχείρηση θα πρέπει να έχουν διάλογο μεταξύ τους και να σέβονται στον άλλο και να μην υπάρχουν επικαλύψεις ε, το, των εντολών τους. Εράχτ, qui j'espère me tiendra pas rigueur d'avoir... Euh, Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θέλω ε, τώρα το λόγο κύριε Έρχαρτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ που με καλέσατε. Raise four points. Very briefly, one a very general one. Um, I think uh, at first we have to ask the question γιατί πρώτα θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι ίδιους, τι συγκρούσεις μας απασχολούν. Ποιο είναι το θέμα μας, διότι έχουμε γίνει μάρτυρες κάποιας αλλαγής και στροφής μετα, από τους βιομηχανικούς πολέμους τους, προς το πολέμους τους εσωτερικούς ε, ή έχουμε την έκφραση πόλεμη των λαών. Εύστοχη, γιατί καλύπτουν αυτό το οποίο έχουμε να επιλύσουμε ως πρόβλημα. Θα πρέπει να δώσει στη τη μάχη για τον λαό πολλές φορές όμως ο λαός που κάθεται και περιμένει να δει την έκβαση. Και άλλο τμήμα του πληθυσμού όμως είναι κατά αυτής τη αντιμετώπισης. Άρα δεν είναι μόνο πόλεμος για το λαό, είναι και πόλεμος κατά του λαού. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ βασικό κοινωνικό πρόβλημα, άρα χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Δηλαδή, έχουμε τώρα μη κρατικούς παράγοντες. Δεν μιλούμε εδώ για κάποια οργάνωση και για ιεραρχία είναι κάτι το πάρα πολύ ρευστό. Πρόκειται για κάποιες συγκρούσεις αέναες. Και είναι αέναες γιατί εδώ δεν γίνεται η σύγκρουση για κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Γι' αυτό το πρέπει τόσο περιβεβλεγμένα. Έχουν αυτούς τους στόχους που τους χαρακτηρίζουμε soft, ευέλικτους. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σφαιρική προσέγγιση. Δεύτερη παρατήρηση. Πρέπει να τονίσουμε τα εξή σημεία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι πολλές δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία. Και όταν δεν υπάρχει τέτοια στιβαρή ηγεσία, υπάρχει πρόβλημα ενότητας. Εγώ δεν είμαι υπέρ της ε, ενότητας της διοίκησης που είναι αδύνατον αυτό, αλλά χρειάζεται ένωση και ενότητα στην προσπάθεια. Άρα χρειάζεται πολιτική ηγεσία επίσης. Δεν έχουμε σε τέτοιου συγκρούσεις ξεκάθαρους στόχους πολιτικούς ή άλλους. Τέτοια είναι η φύση αυτής της ε, σύγκρουσης. Πολλές φορές επομένω είναι πρόβλημα συντονισμού και επίσης αφού μιλούμε για σύγκρουση κατά την οποία έχουμε ανασυγκρότηση παράλληλα με τον πόλεμο, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τι θα πρέπει να κάνει κανείς. Μερικοί λένε να γίνουν και τα δύο, ταυτόχρονα. Ανασυγκρότηση και μάχη. Εκεί, στον τόπο της μάχης. Όχι, άλλοι λένε ότι θα πρέπει η ανασυγκρότηση να γίνει εκτός των πεδίων μαχών. Κάτι άλλο τώρα. Να, ισχύει για το Αφγανιστάν. Πώς κανείς θα πείσει κάποιους που τους έχει παραμιλήσει επί μια εξαιτία επτά αιτία. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί. Ιδίω όταν έρθει η ώρα να ετοιμαστεί μια καινούργια αποστολή. Άλλο, έβδομο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο ήδη το ανέφερε κάποιος από τους ε, προλαλήσαντες. Δεν έχουμε αρκετές ε, πληροφορίες για την επιτόπου κατάσταση. Χρειάζεται να έχουμε περισσότερη, περισσότερη πληροφόρηση για το τι επικρατεί σε κάθε χώρα και αυτό να, γίνεται από τους ε, συνομιλητές μας, τους επιτόπου, τους τοπικούς, τους ντόπιου. Άρα θα πρέπει να ζητάμε τους σωστούς συνομιλητές. και ο σημερινό φιλός αύριο μπορεί να γίνει εχθρό. εδώ πέρα για το θέμα τώρα της διαφθοράς. και η κυβέρνηση που καλείται να αποφασίσει αν πάει τις του κράτους στα χέρια της. Από την άλλη μεριά θα πρέπει και εμείς να δούμε ανάλογα με το πόσο η ηθική κυριότητα έχουν αυτοί, τι προσέγγιση θα υιοθετήσουμε. Third point, what does this mean for a comprehensive approach? I think the first lesson is, or the first... Τώρα, τι πώς του διευθυντή κανείς, μου, γιατί μια σύσταση θα μπορούσε να είναι ότι ο πάντοτε θα πρέπει να έχει μετά του οίκου του σφαιρική αντιμετώπιση. Γιατί αν κανεί δεν μπορεί να έχει τέτοια σφαιρική αντιμετώπιση προ τα μέσα, τότε δεν μπορεί να τα κάνει ούτε σε προ τα έξω. Κατά δεύτερο λόγο. Δεν θα πρέπει κανεί ποτέ να ξεχνά ότι υπάρχουν ένα σωρό φραγμοί και εμπόδια, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει με τέτοιου είδου ε, έκτακτε καταστάσει. Φραγμοί όσον αφορά την πολιτική, όσον αφορά την συνεργασία του με κάποιους ε, εμπλεκόμενους και δεν μιλάμε τους ομιλίε μόνο στην ε, χώρα εκείνη, γιατί υπάρχουν και εκεί πέρα πολλέ παρεξηγήσει. Στη χώρα επέμβαση επίση είναι πάρα πολύ βασικό το να υπάρχει μια βαθιά ανάλυση κατάστασης, να ξέρει κανείς με ποιον έχει να κάνει, θα πρέπει επομένως κανείς να ξέρει σε βάθος την κοινωνία στην οποία απευθύνεται, να ξέρει κανείς από τι ταλανίζεται αυτή η κοινωνία. Τέτοια προσέγγιση χρειάζεται. Ας την πούμε στρατηγική. Κάτι άλλο τώρα. Θα πρέπει κανείς να κάνει τις σωστές υποθέσεις και όχι τις λάθος. Ανάπτυξη, σταθερότητα. Πώς συνδέονται αυτά. Είναι το ένα φυσική συνέχεια του άλλου, φυσική συνέπεια του άλλου. Μα είναι δυνατόν η φτώχεια να θεωρείται ότι είναι η υποχρεωτική αφετηρία της σύγκρουσης. τέτοιου είδου ερωτήματα πρέπει να θέσει και να τα θέσει σωστά. Φυσικά θα πρέπει να, να, να κοιτάξει και τα του πολιτικού προσωπικού, όπω ήδη ενεφέρθηκε. Εδώ πέρα έχουμε ένα κενό ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων, αλλά αυτό αφορά κάθε δραστηριότητα. Παντού και επί το θα πρέπει κανένα να επενδύσει περισσότερο στι δυνατότητε του πολιτικού προσωπικού. και άλλο το οποίο πρέπει να σας πω δύο λίγο και το οποίο είναι ότι θα πρέπει κανείς να σέβεται την εντολή των άλλων εμπλεκομένων και το οποίο ήδη μας ανέφερε η συνάδελφος. Τέλος, να μην θεωρείτε ότι όλα είναι δυνατόν να τα κάνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θα πρέπει κανείς να ξέρει ποια είναι τα όρια. Τα όρια κάποιου που είναι έξω από το χώρο. Τι μπορεί να πετύχει σε μια χώρα όπου το περιβάλλον είναι εχθρικό. Τι σημαίνει όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέντε συμπεράσματα. Πρώτα πρώτα. Προσοχή με οποιαδήποτε εμπλοκή. Δεύτερον. Αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού και ένταξή του στην στρατηγική. Τρίτον. Ε, εμπειρογνωμοσύνη και ανάλυση της κατάστασης. Εξέταση εναλλακτικών λύσεων από think tanks, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από ειδικού, οι οποίοι να είναι ντόπια. Πάρα πολύ βασικά όλο αυτό. Τέταρτον. Θα πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ βαθιά όσον αφορά την πολιτική λύση πριν την εμπλοκή. Και μην ξεχνά κανεί ότι μπορεί να καταφέρει μόνο όσο είναι δυνατόν να κάνει για να συνεισφέρει στην λύση του προβλήματος, γιατί το πρόβλημα καταρχήν συνδέεται με αυτή τη χώρα και με τον λαό, τον εμπλεκόμενο που τον αφορά. Άρα θα πρέπει, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη οποιαδήποτε λύση προς συμμετοχικές στατικές. Δεν υπάρχει καμία πανάκια. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχία. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε το έλασον κακόν, αλλά χωρίς όμως σφαιρική προσέγγιση πάλι δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Επομένως, ποια είναι η ελλακτική λύση, μόνο δύο βλέπω. Μη εμπλοκή και δεύτερον, πάρα πολύ πρώιμη εμπλοκή, σαν πρόληψη. Αν όμως φτάσουμε στην εμπλοκή, σε εχθρικό περιβάλλον, θα πρέπει αυτό να γίνει με τα λόγου γνώσεως, ξέροντας ότι κανείς θα πρέπει να αφοσιωμένος ολόψυχα, στο στρατηγικό στόχο και όχι μόνο στην τακτική. Merci, Monsieur Dear Chairman, dear ladies. Uh, ε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την άποψη να παρουσιάσω τις ιδέες μου σε αυτό το διακεκριμένο ακροατήριο. Θα αναφερθώ στις τάσεις της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, στη βάση της εμπειρίας και των γνώσεων που, των συγγραφέων του έργου ε, το οποίο αποτελείται από έξι κεφάλαια που αφορούν τα διέξοδα και τις τάσεις. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω το εξής. Ε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες σε πολλαπλά επίπεδα. Όλοι θεωρούν ότι ένας πετυχημένος συντονισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη σταθεροποίηση. Οι δυσχέρειες ε, ανακύπτουν όταν πρέπει κανείς να ορίσει ποιος είναι ακριβώς ο συντονιστής και τι θα πρέπει να συντονίσει. Γιατί όλοι θέλουν να συντονίσουν, αλλά κανείς δεν θέλει να είναι αντικείμενο συντονισμού. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχές πολιτικο-στρατιωτική συνεργασία, ορισμένε ανθρωπιστικέ ε, ενώσει δεν θέλουν να συνεργαστούν με στρατιωτικές δυνάμεις, φοβόμενοι θα χάσουν την ε, ουδετερότητά τους. Ε, ορισμένες ανθρωπιστικές ενώσεις, από την άλλη, είναι, έχουν πολύ πιο πραγματιστικό προσανατολισμό και μπορούν να συνεργαστούν με στρατιωτικές δυνάμεις. Όσον αφορά τον τοπικό πληθυσμό, ε, δεν γνωρίζουν πάντοτε ποιος θα τους παράσχει συνδρομή. Ορισμένοι ε, πολίτες εκπλήσονται να διαπιστώσουν ότι υπάρχει μία αντιπαράθεση όσον αφορά το στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σκέλος και ορισμένοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί ε, συμμετέχουν σε ανοικοδόμηση. Στο Αφγανιστάν η έρευνα δείχνει ότι ε, πολλοί ε, εμπλέκονται σε τέτοιου είδους αδιέξοδα. Ε, το άλλο πρόβλημα είναι η πληθώρα των παραγόντων. Ε, υπάρχουν ε, εκατοντάδες μη κυβερνητικών ενώσεων. Μόνο στη Σρι Λάνκα μετά το τσουνάμι ε, υπήρξαν χιλιάδες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Το ίδιο ισχύει και για στρατιωτικές ομάδες, όπου, τον οποίο ο αριθμός ποικίλει σημαντικά. Για παράδειγμα, στο Αφγανιστάν υπάρχουν, έχουν αναπτυχθεί ε, στρατιωτικές ε, δυνάμεις από διάφορες ε, χώρες και οι ίδιες αποτελούνται από πάρα πολλά τμήματα. Κάτι το οποίο περιπλέκει εξαιρετικά τα πράγματα, καθώς και η διαπλοκή τους με τον τοπικό πληθυσμό και Τέλος, όχι μόνο ο αριθμός των ομάδων, αλλά και πάρα πολλές ε, μη στρατιωτικές ε, ομάδες ε, ανήκουν σε διάφορα επίπεδα ιεραρχίας. Ένας επαρκής συντονισμός όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ όλων αυτών των διαφορετικών επιπέδων οδηγούν σε πάρα πολλές συγκρούσεις. Στο Κονγκό η σημασία της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας έχει διαπιστωθεί τοπικά, αλλά ο συντονισμός της ε, πολιτικής στη Κινσάσα εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών ε, είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. Ε, και πολλές φορές γίνεται από την κάρτα στη Βιέννη, για παράδειγμα, ένα συντονισμός, κάτι το οποίο είναι, δεν μπορεί να είναι τελέσφορο. Υπάρχουν στις διάφορες αυτές ομάδες διαφορετικές ερθωτικές δομές και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Ε, το στατικό σκέλος, οι μη κυβερνητικέ ε, ομάδες ε, θέτουν εντελώς διαφορετικές απαιτήσει. δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μία ενιαία προσέγγιση γιατί υπάρχουν ε, διάφοροι εκπρόσωποι που διαθέτουν ε, ελλειπείς ε, πληροφορίες. In engaging members... Όσον αφορά τις αποστολές, κάποια μέλη της Εθνούς Κοινότητας ε, μετέβησαν σε απομακρυσμένες περιοχές προσπαθώντας να μελετήσουν την ποιότητα της προσφοράς και τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνεται κείμενο διαχείρισης μια δράση. Πολλές ε, φορές ε, οι επιχειρήσεις αυτές είναι συνάρτηση της επιτόπιας ε, ζήτησης. Και... Αλλά θα πρέπει αντί να υπακούν σε διεθνείς κανόνες. Υπάρχει μία αυθαιρεσία όσον αφορά την εφαρμογή αξιών ή κανόνων. Υπάρχουν κάποιοι εγχώροι παράγοντες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές και αυτό μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους και να αυξήσει το βαθμό ασφαλείας. Η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων επίσης μπορεί να μειώσει το χάσμα μεταξύ τοπικών κοινοτήτων και εξωτερικής παρέμβασης, ε, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικοδόμηση της ειρήνης. Με αυτό μειώνεται το χάσμα όσων μεταξύ τοπικών και μη τοπικών παραγόντων και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται μακροπρόθεσμα η αποτελεσματικότητα της αποστολής. Όσον αφορά την τοπική συμμετοχή στην Αφγανιστάν, εδώ μπορείτε να δείτε τις ε, κατευθυντήριες ε, γραμμές που διέπουν ε, την συμπεριφορά των ομάδων του ειδικού εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών και των εκπροσώπων, των άλλων εκπροσώπων του ΝΑΤΟ. Ε, πουθενά σε όλα αυτά δεν αναφέρεται η συμμετοχή των ε, τοπικών παραγόντων. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για την τρέχουσα κατάσταση. Τώρα, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα όσον αφορά το επίπεδο της κατάρτισης. Ε, αφού οι πόλεμοι στην Ευρώπη οδηγήθηκαν σε ένα τέλος, μόνο ε, το ΝΑΤΟ δημιούργησε τα δικά του δόγματα για πολιτικοστρατηγική συνεργασία. Στη Βοσνία και στο Κόσοβο, τα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορέσαν να αναπτύξουν ε, ε δυνάμεις με επαρκή κατάρτιση υπάρχουν, υπήρξαν σοβαρά ε, ελλείμματα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και έτσι ήταν μειωμένη η συμβολή στην προσπάθεια νοικοδόμησης της χώρας. Για να απαλληφθούν αυτές οι διαφορές θα πρέπει η υπάλληλοι που ασχολούνται με ανθρωπιστικά θέματα να είναι ενήμεροι για ζητήματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί να είναι ενήμεροι για θέματα ανθρωπιστικής συνδρομής. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνειδητοποίηση όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους. Και οι διαφορές αυτές θα πρέπει να τονίζονται ήδη κατά την ε, ε, εκπαίδευση. η πολιτικοστατική συνεργασία είναι ένα θέμα το οποίο δεν λαμβάνεται πολλές φορές ε, σοβαρά υπόψη. Στην ε, Ακαδημία Άμυνα, της Ολλανδίας ε, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ζητήματα πολιτικοστατικής συνεργασίας και νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Ορισμένες οργανώσεις παρέχουν ολοκληρωμένα μαθήματα και το ΝΑΤΟ παρέχει ολοκληρωμένα μαθήματα όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού. Ορισμένες στρατιωτικές ε, δυνάμεις ε, εισήγαγαν αυτά τα μαθήματα ούτω ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Είναι σημαντικό για να μην υπάρχει και επικάλυψη με προηγούμενες δραστηριότητες. είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέχεια. Ένα τμήμα της εκμάθησης γίνεται και επί τόπου. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ορισμένων μιας στρατιωτικής πλατφόρμας, ούτως ώστε να αυξηθεί η συγκέντρωση πληροφοριών κατά τη φάση της ανάπτυξης των δυνάμεων. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να αντλούνται και τα διδάγματα από όλα τα, αυτά τα μαθήματα. Και θα πρέπει να υπάρχει μια πλατιά ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κυβερνήσεων μετά τις ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ορισμένες από τις ε, πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές τις ε, ασκήσεις είναι θεμελιώδη σημασία. Και θα πρέπει να υπάρχει μια ανταλλαγή όσον αφορά τα διδάγματα που μπορούν να αντιληφθούν από προηγούμενες επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των μελλοντικών ε, δράσεων. Η πρόκληση είναι να εξασφαλίσει κανείς ότι αξιοποιείται η εμπειρία για τις μελλοντικές αποστολές και εντάσσεται στα μαθήματα εκπαίδευσης και άσκησης. Ε, η θεωρία και η πρακτική θα πρέπει να είναι αλληλένδετες και θα πρέπει να γίνει μια εις ε, έρευνα όσον αφορά την πολιτιστική συνεργασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Et enfin, Monsieur Richard Wright, qui nous a rejoint que je salue directeur à la DG Rolex de la Commission. Chairman uh, Donjon, um, ladies and gentlemen, thank you very much, first of all, for... Πρόεδρε Ντανζόν, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την πρόσκλησή σα και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να ακούσω όλε τι παρουσιάσει. Μόλι έρχομαι από μια ε, συνεδρίαση του Συμβουλίου και δεν μπόρεσα να έρθω στην ώρα μου. Αλλά θα ήθελα να σχολιάσω ένα-δυο από τα στοιχεία που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και με τους Υπουργούς Αμήνης, γιατί είναι σχετικά με τη σημερινή συζήτηση. Να ξεκινήσω τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει έναν βασικό ρόλο στη διαχείριση κρίσεων και στην ε, συνεργα... πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Και φυσικά ο ρόλος αυτός θα αλλάξει όταν θα έχουμε την υπηρεσία εξωτερικών... εξωτερικής δράσης, αλλά να θυμίσω κάποια σημεία κλειδιά που θα ισχύσουν και θα συμβάλλουν στην προσπάθεια της Ένωσης. Ε, παραδοσιακά μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια, προστασία μάχων μέσα σε περιβάλλον κρίσης. Επίσης έχουμε μια, ένα μέσο ταχείας αντίδρασης, ένα βραχυπρόθεσμο αλλά και, βραχυπρόθεσμο, και μακροπρόθεσμο ε, στοιχείο που μας βοηθά να φτιάξουμε ένα στοιχείο αντίσταση στις διαπεριφερειακές απειλές. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ε, φτιάχνουμε ε, εταιρικέ σχέσεις με τις ΜΚΟ για την οικοδόμηση ειρήνης, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργαζόμαστε γι' αυτό. Να τονίσω επίσης πως πάντοτε πάντοτε συνεργάζεται στενά και το υπογραμμίζω αυτό με τις αποστολές CSTP, είτε αυτές είναι στρατιωτικής είτε είναι πολιτικής φύσης. Να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα. η στρατιωτική αποστολή του Τσάντ που τώρα έχει περάσει στις, στον ΟΗΕ ήταν ένα καλό παράδειγμα ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση κρίσεων είχαμε από τη μια πλευρά είχαμε 300.000 στρατιώτες που προστάτευαν τα στρατόπεδα των ε, εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων στο ανατολικό Τσάντ Ταυτόχρονα είχαμε σημαντικά ανθρωπιστικά και βοήθεια και αναπτυξική βοήθεια που δινόταν στους πρόσφυγες στα στρατόπεδα και επιπλέον χρησιμοποιώντας το μέσο σταθερότητας με τις ε, διατάξεις του για την ανταπόκριση σε μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε τον ΟΗΕ που παρήχε ε, εκπαίδευση στην αστυνομία του Τσάντα αλλά και προληπτικές δράσεις. Πολύ καλό παράδειγμα συνδυασμού όλων των διαθέσιμων μέσων για να επιτύχουμε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Να τονίσω επίσης ένα άλλο παράδειγμα στη Γεωργία. Αυτή τη φορά στον πολιτικό τομέα, σε ανταπόκριση στην κρίση του 2008 και στην εγκαθίδρυση μιας ευρωπαϊκής αποστολής παρακολούθησης πολύ γρήγορα το Σεπτέμβριο, μέσα σε 17 μέρες. Και να ανοίξω μάλιστα μια παρένθεση, πως δεν πιστεύω πως οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός θα μπορούσε να φτιάξει μια τέτοια ε, αποστολή τόσο σύντομα και ήταν θαύμα πώς τα κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν έδωσε σημαντική βοήθεια και ακολουθήθηκε αμέσως μια μεγάλη διάσκεψη δωρητών για τη Γεωργία και πάλι όλα αυτά έγιναν μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής πολιτικής ιδέας. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο για, σε μια κοινή ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικοστατικής συνεργασίας, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, καλύτερα, με μεγαλύτερη συνέπεια και αυτό νομίζω θα το καταφέρουμε όταν θα φτιαχτεί Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία που σήμερα συζητήθηκε και πάλι στη Λουξεμβούργο. Από τη δική μου προοπτική και είμαι σίγουρο ότι ο συνάδελφο Διντιέ Λενουάρ θα έχει πει τα ίδια νωρίτερα. Εμεί ξεκινάμε από την αρχή τη ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό ε, αναφέρεται σαφώς στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια του 2003, εφαρμογή της οποίας εξετάστηκε στα τέλη του 2008 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Προεδρίας και νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Κομισιόν είναι η σαφής δήλωση ότι η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι θεμελιώδης σημασίας, θεμελιώδης σημασίας και πρέπει, είναι αλληλένδετα και θα πρέπει και τα δύο να αντιμετωπίζονται όταν έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις κρίσης και βάσει αυτής ε, της γραμμής προχωράμε και νομίζω ότι όλα είναι και περισσότερα παραδείγματα έχουμε για το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Να στραφώ σε ένα-δυο τομεί που συζητήθηκαν σήμερα στο Συμβούλιο. Καταλαβαίνουμε ότι σα διανέμονται και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Α δούμε το Αφγανιστάν. Είμαι σίγουρο πως το έχετε ήδη αναφέρει. Στο Αφγανιστάν έχουμε μια κατάσταση όπου προφανώς υπάρχει ένα πολύ έντονο συντηρητικό στοιχείο, ISAF NATO, ε, την, ταυτόχρονα έχουμε μεγάλη εμπλοκή της Ένωσης μέσω της ε, αποστολής της αστυνομικής, της UPOL, και θα, καταλάβα, θα έχετε καταλάβει και από την πλευρά του ΝΑΤΟ και από την πλευρά της Ένωσης ότι συλλογικά πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των ε, αφγανικών ε, ε, δυνάμεων ασφαλείας, δηλαδή αστυνομία και ένα είδος αστυνομίας ζαντάρμα, τύπου ζαντάρμα. Κανένα μέρος δεν μπορεί να τα καταφέρει αυτά όλα μόνο του. Πρέπει να υπάρξει γενικά συνεργασία. Έχουμε να αναπτύξει ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα δράσης στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε σε επίπεδο ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και άλλο ένα στοιχείο που θέλω εδώ να τονίσω είναι η ανάγκη η χρηματοδότηση να διαχειτεύεται μέσω της κυβέρνησης ε, του Αφγανιστάν. Μια από τις προκλήσεις είναι ότι ε, η χρηματοδότηση προς το Αφγανιστάν δεν περνά από το κυβέρνηση και άρα λοιπόν και πρέπει να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή η μας είναι να διοχετεύεται η χρηματοδότηση όλο ένα και περισσότερο μέσω τη κυβέρνηση. Το πρόγραμμα δράσης της Ένωση δεν καλύπτει όλη την βοήθεια προς το Αφγανιστάν. Μίλα μόνο για το τομεί όπου θα εστιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το σχέδιο τώρα καθοδηγείται από την πρέσβυρα, τον πρέσβη μάλλον, ε, ειδικό εκπρόσωπο, πρώην ε, Υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας. Ελπίζουμε πως θα προωθήσει αυτό τη δική μας ε, θέση στην χώρα. πολύ, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. είμαι σίγουρος ότι θα αναφέρθηκαν και οι αποστολές της Σομαλίας την οποία διαχειρίζεται τη Διέ Λενουάρ και οι συναδελφοί του, αλλά και πάλι όλα αυτά τονίζουν ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Η αποστολή μας ήταν επιτυχής, βοήθησε στο να περιοριστούν τα περιστατικά πειρατείας. Ακόμα όμως αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα ενός προβλήματος, όχι τα αίτια. Και γι' αυτό χρειάζεται κοινή προσπάθεια ώστε να ενισχυθούν οι θεσμοί στη Σομαλία. Μια μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και πάλι καταβάλλονται προσπάθειες από την Ένωση για να εκπαιδευτούν υπηρεσίε ασφαλείας που θα <clears throat> υπηρετήσουν αυτή την κυβέρνηση. Αλλά πρέπει να διεξασφαλίσουμε ότι αυτές οι δυνάμεις θα πληρώνονται καθώς και την προσπάθειά μας στην ανθρωπιστική βοήθεια αναπτυξιακή βοήθεια, να ενισχύσουμε τις θαλάσσιες δυνατότητες των χωρών στην περιοχή και να στηρίξουμε όλα τα κράτη εκεί ώστε να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Έχουμε συμφωνήσει κάποιες ε, συμφωνίες σε μεταφοράς με κάποια κράτη. Θέλουμε να προωθήσουμε περιφερειακή προσέγγιση στο πρόβλημα, αυτό είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα επιθυμεί να προωθήσει η ΠΑΤΟΣ εκπρόσωπος ε, για τη χρήση των τοπικών ε, οργανώσεων. Ας στραφώ τώρα σε έναν άλλο τομέα πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας, όπου στο θαλάσσιο τομέα και στο τομέα της θαλάσσιας εποπτείας, πράγμα που συζητήθηκε από τους Υπουργούς Αμήνες σήμερα. Η θαλάσσια εποπτεία καταρχήν είναι πολιτικό ζήτημα, γιατί 90% των πληροφοριών εποπτείας προέρχεται από τον πολιτικό τομέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που ηγείται εδώ και προτιμάζει αυτό που λέμε ένα περιβάλλον, ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανταλλαγή πληροφοριών. Προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς, μπορεί να είναι ευρωπαϊκές υπηρεσίες, αλλά είναι και υπηρεσίες των κρατών μελών και στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχουν αρκετές τέτοιες υπηρεσίες. Αλλά επίσης αυτό σημαίνει συνεργασία στενή με τη στρατιωτική πλευρά και με το ναυτικό, τις ναυτικές δυνάμεις των χωρών. Γενικό γενικός μας στόχος είναι να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς για την αυσιπλοεία να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να μπορούν να διεξάγουν τις δραστηριότητε τους. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προωθεί το στόχο της σύστασης ενός προγράμματος δράσης, προγράμματος εργασίας, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Συμβουλίου. Σήμερα, στην συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Αμήνης, ένα από τα συμπεράσματα καλεί την Κομισιόν καθώς και τη Γραμματεία του Συμβουλίου και τα κράτη-μέλη, να εξετάσουν κατά πόσο μπορούν να διερευνήσουν επιλογές ώστε να αναπτυχθεί μία ε, στρατηγική ασφάλεια στην αυσιπλοεία μέσα στο πλαίσιο της CFTP. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε άλλο ένα παράδειγμα όπου υπάρχει επικάλυψη των προσπαθειών πολιτικής και στρατιωτική και τα δύο θα πρέπει να συνδυαστούν ώστε να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή καλύτερη ναι, εποπτεία στην αυσιπλοεία. Έγινε συζήτηση για το πώς θα συνδυαστούν καλύτερα οι δυνατότητες που έχουμε για την αποφυγή θαλάσσιων καταστροφών μετά από την, ε, ή για επίγουσα βοήθεια όπως μετά από την εμπειρία της ΑΕΤΗΣ, πώς θα ενισχυθούν δηλαδή οι δυνατότητες ε, πολιτικοσυνδετικές και στον ερευνητικό τομέα. Όταν κανείς λοιπόν συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία και από την επιχειρησιακή πλευρά και το τι κάνουμε από την πλευρά των δυνατοτήτων, αυτό το οποίο προκύπτει είναι μια διάσταση μεγάλη έντονη συνεργασία, δηλαδή είναι ανάγκη ο συνδυασμό των δύο και η συνεργασία μεταξύ των δύο. Τέλος, να συμφωνήσω με έναν από τους προηγούμενους ομιλητές που άκουσα, ότι δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης και αυτό είναι αλήθεια. Πολύ δουλειά γίνεται σε αυτούς τους τομείς και σίγουρα και στο μέλλον θα γίνει παρόμοια προσπάθεια και στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης αλλά και στον ΩΣΑ και στην Επιτροπή προσπαθούμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις δυνατότητες πρόληψης των συγκρούσεων. Είναι πολύ σημαντική πτυχή. Από τη στιγμή που ξεκινάνε οι συγκρούσεις, το κόστος για όλους είναι πολύ μεγαλύτερο από, την πρόληψη, από το κόστος της πρόληψης. Πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για το μέλλον, άρα επ' αυτού θα πρέπει να εργαστούμε. Και σε αυτά, με αυτά θα κλείσω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία απευθύνεται προς τον κύριο Ράιτ που μόλις μίλησε και είναι εξής. Θα ήθελα ακριβώς εν ώψη της αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, θα ήθελα να ακούσω ότι ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε θα μπορούσε να είναι ε, δεσμεύσεις που αναλαμβάνει κανείς, ε, θα πρέπει να τις εκπληρώνει. Δυστυχώς δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Και διαβάζοντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Συμβουλίου που μόλις έχουν ε, διανεμηθεί, Υπάρχουν εδώ τρεις ε, παράγραφοι για την πόλη στο Αφγανιστάν και σε καμία από αυτές τις παραγράφους δεν αναφέρεται καν η προοπτική η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010 να προσπαθήσει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά το ε, μέγεθος των ε, δυνάμεων εκεί. Και νομίζω ανάψε όλων αυτών η συζήτηση αυτή ε, εμφανίζεται γελία εδώ. Θα μπορεί, μπορεί να σορθοκομιλίζει κανείς. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά που ακούσαμε προηγουμένως είναι μία προσπάθεια α, στρουθοκαμιλισμού ή ψεμάτων ε, εξέροντας τις ε, προσπάθειες της Ιουπόλ e χωρίς να ομολογεί κανείς το γεγονός ότι είναι όνειδος ότι η UPOL ε, βρίσκεται, κινείται πολύ χαμηλότερα από το, ευκταίο, από το υποσχεθέν ε, επίπεδο. Ε, το δεύτερο ερώτημα αφορά τον κύριο Ρίτιενς από την Ολλανδική Ακαδημία Άμυνας. Αν κατάλαβα καλά τα όσα είπατε, κύριε Ρίτιενς, είπατε ότι στο Αφγανιστάν ο εγχώριος πληθυσμός αδιαφορεί για το, την πηγή της ε, βοήθειας ε, και δεν μπορούν καν να καταλάβουν αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα ήθελα να σε επισημάνω μία δήλωση του Προέδρου της Ένωσης των αναπτυξιακών μη κυβερνητικών οργανισμών, Γιώργεν Λίζε, ο οποίος σε σχέση με το θέμα αυτό είπε τα εξή και παραθέτω το απόσπασμα. Υπάρχει μία ατυχής ε, σύγχυση των ορίων αρμοδιοτήτων μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων και ανθρωπιστικής ε, εντολής και πολιτικών ε, μη στρατιωτικών οργανισμών που θα πρέπει να είναι ουδέτερες. Τέλος του παραθέματος. Και θα ήθελα να φέρω και μία δήλωση του Αντιπροδέδρου Ζακ Φώστερ της CIFC και το λέω στα αγγλικά. Ο βασικός κίνδυνος της ανθρωπιστικής ε, δράσης είναι η ένταξή του στην ε, πολιτικοστρατηγική στρατηγική για να νικήσει τον εχθρό. Με άλλα λόγια, η υπαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων σε πολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας τα σαν ένα εργαλείο για την ε, τοπική πολιτική. Οι ανάγκες του πληθυσμού είναι να θεωρήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια σαν ένα εργαλείο ξένης ε, παρέμβασης. Θα ήθελα να σχολιάσετε σχετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς τον κύριο Ρίτκινς και χαίρομαι πάρα πολύ που μπόρεσε να έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το ερώτημά μου σχετίζεται με το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Μπίτι Κόφερ. Εάν σε ένα στρατικό θέατρο, μια στρατική σκηνή, οι μη στρατικές δυνάμεις δεν λειτουργούν πλέον και στην περίπτωση αυτή οι Αφγανές, αφγανικές ε, πολιτικές ε, οργανώσεις. Έχουμε μια έλλειψη μη κυβερνητικών οργανισμών ή οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί ε, λόγω οικονομικών περιορισμών δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως. Αληθεύει ότι οι δυνάμη, δυνάμεις θα πρέπει να έχουν τεχνογνωσία και, την, και τις ικανότητες στο πολιτικό επίπεδο, στο μη στρατιωτικό επίπεδο, δηλαδή πώς μπορούν να προωθήσουν την οικονομία, να ξαναφτιάξουν τους δρόμους κλπ. Δηλαδή, όχι στενά στρατιωτικέ λειτουργίες. Κάτι το οποίο όμως ενδεχομένω θα είναι αναγκαίο γιατί κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Και ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε στην περίπτωση αυτή από την περίπτωση του Αφγανιστάν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την κυρία Κρίλ. Η ανθρωπιστική βοήθεια καμιά φορά ε, εγκυμονεί κάποιου κινδύνου. Υπάρχουν ε, πολλοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί που εργάζονται χωρίς καμία μορφή κάλυψης ή ασφάλειας. Γι' αυτό ε, πολλές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το φέδρο του πολέμου. Η δική σας οργάνωση οργανώνει κάποια τμήματα κατάρτισης ή προπαρασκευής για να παρακαμφθούν, για να ξεπεραστούν ακριβώς οι κίνδυνοι των εθελοντών που δουλεύουν εκεί. Ε, ναι, και εγώ είχα προετοιμάσει το ίδιο απόσπασμα όπω ο κύριος Μπιουτικόφερ, το ίδιο παράθεμα. Και πραγματικά θα ήθελα να μου απαντήσετε ένα ανάλογο ερώτημα. Η κυρία Κρίλ παρουσίασε αντίστοιχα τα πράγματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πτυχή και νομίζω και το κύριο Ρίτχενς το είπε. Είπατε ότι θα πρέπει να συμμετέχει και η χώρα υποδοχής. Το είπα ήδη πριν από μία ώρα ότι θα πρέπει να εμπλακούν οι τοπικές δομές, να συμπεριληφθούν οι τοπικές ιδιομορφίες. Ωστόσο, ε, ο στρατός ε, εξορισμού έχει έναν πατριαρχικό προσανατολισμό και είναι αδιάφορο αν υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών. Η δομή του στρατιωτικού είναι πατριαρχική και ιεραρχική. Οι γυναίκες φοβούνται τους στρατιώτες, οι γυναίκες φοβούνται το στρατό και αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Και νομίζω ότι αυτό ότι είναι σε απόλυτη αντίφαση το να λέμε ότι οι στρατιωτικοί είναι σε θέση σε μια Ισλαμική χώρα, για παράδειγμα όπω είναι το Αφγανιστάν ή στην Αϊτή, πραγματικά να συμπεριλάβουν τι ενδότητε των γυναικών στη δικασία επίλυση των συγκρούσεων. Όπω είπε η κυρία Λούνετσεκ, ε, φαντάζομαι ότι οι δυνατότητε των γυναικών είναι, πηγαίνουν πολύ πιο πέρα από το να αποκαλύψουν που κρύβουν ε, οι άντρες τα όπλα τους. Αναφέρατε αυτό το παράδειγμα, κυρία Λούνατσεκ. Ε, θα ήθελα να σε επισημάνω ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ε, λειτουργίες των γυναικών εντός μιας κοινωνίας που δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν από τους οδητικούς. Ε, κύριε Ρίτιενς, ε, μιλήσατε, για, αναφερθήκατε στα παιχνίδια ρόλων και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια μοιραία πτυχή των, ε, του παιχνιδιού αυτών των ρόλων, στο Κωσφοπαίδιο. Εκεί η πολιτικο συνεργασία, ειδικά μεταξύ της Γιούλεξ και του ε, ΝΑΤΟ, λόγω πολλών ε, διαδηλώσεων γίνεται η προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι διαδηλωτές. Ε, έγιναν ε, στους τελευταίους μήνες ε, τρεις τέτοιες ασκήσεις και το, που βασίζονται ακριβώς σε τέτοια παιχνίδια ρόλων και το περιεχόμενο μιας τέτοιας άσκησης βασιζόταν σε ένα σενάριο όπου λόγω του επικείμενου ε, κλεισίματος ενός ε, νοσοκομείου ε, γίνονταν διαδηλώσεις των εργαζόμενων σε αυτό το νοσοκομείο. Και ακριβώς η, στην άσκηση αυτή συμμετείχαν και οι πολιτικές δυνάμεις, κάτι το οποίο θεωρώ τελείως παρά, απαράδεκτο, θεωρώ άστοχο ένα τέτοιο, μια τέτοιου είδους άσκηση, πολιτικο-στρατιωτική άσκηση. Το πώς να πατάξει κανείς δηλαδή τις διαδηλώσεις εργαζόμενων σε ένα νοσοκομείο θα έλεγα ότι στο μέλλον θα πρέπει να γίνουν προσεκτικές αναλύσεις όχι μόνο των επιτόπιων προβλημάτων μιας χώρας, αλλά επίσης θα πρέπει να γίνουν εμπεριστατωμένες και προσεκτικές αναλύσεις εν σχέση με τα συμφέροντα ορισμένων χωρών που επιθυμούν να συνεχίσουν τη συνεργασία ε, τέτοιων κυβερνήσεων όπως στο Κονγκό και τους εξοπλίζουν με όπλα και βοηθούν στην ενίσχυση των ε, στρατών, ε, στρατοί που εξαπολύουν ολέφρεις επιθέσεις κατά των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Για το, για το Κόσοβο τώρα. Όσον αφορά την τρίτη της τάξης, ε, πολλές φορές έχουν ξεπεραστεί όλα τα σενάρια από την πραγματικότητα. Στη Μητρόβιτσα, ε, πριν από λίγους μήνες έγιναν κάποιες διαδηλώσεις και ε, οι διαδηλωτές είχαν ε, όπλα, ήταν όπλα Είχαμε Ουκρανούς και Γάλλους στρατιώτες του ΟΙα, που έχασαν τη ζωή τους και τις δύναμεις παρεμβολής. Οπότε πάρα πολλές φορές δεν είναι καθόλου ειρηνευτικές αυτές οι διαδηλώσεις. Κύριε Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις προς τον κύριο Ράιτ. Ήρθα αυτό μας είπατε στο Τσάδα. Είπατε πάρα πολύ καλό παράδειγμα ολοκληρωμένης προσέγγισης. Το προηγούμενο πάνελ ακούσαμε τον κύριο ότι προσπαθήσατε εκεί να έχετε τέτοια προσέγγιση. Και όντω κάτι καταφέρατε σε αυτή την προστασία τη ζωή, αλλά από πλευρά πολιτική ή στρατιωτική δεν μπορείτε να πείτε ότι ήταν επιτυχημένη η αποστολή. Η ε, κυρία Κρύλ επίση αναφέρθηκε ότι απέτυχε αποστολή. Εσείς είπατε ότι πέτυχε. Έχουμε επομένω εδώ διαφορετικέ απόψεις. Υπάρχει κάποια παρεμβολή ε, και δεν ακούγεται η ομιλήτρια. Νομίζω ότι θα αποδώσει αυτή η προσέγγιση. Ή μήπω ήταν ε, το θέμα η μηπω ηταν το θεμα η να το μελλον για το ποιο ρόλο θα παίξει η Γαλλία κλπ. Επομένω, είναι τα πρώτα συμπεράσματα από το πρώτο πάνελ που τουλάχιστον εγώ συγκράτησα είναι ότι έχουμε αυτή την έλλειψη κοινού πολιτικού στόχου. Αυτό ήταν ε, το επιζήμιο για αυτές τις κοινέ αποστολέ. Για πέστε μου τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Επίσης, γιατί Γιούλεξ, στο Κόσοβο. Διαβάζω τα συμπεράσματα τα σημερινά του Συμβουλίου και αναφέρεται ότι για να θα πάω στο Συμβούλιο σε τέσσερις μέσα ανησυχήτρια. Λέει λοιπόν για το πώς σήμερα ενεργεί η Γιούλεξ. Τι κάνει και τι δεν κάνει. Και αναφέρονται όλα αυτά, όπως και λέει επίση όσον αφορά την εκδίκαση κάποιων πάρα πολύ δύσκολων ποινικών υποθέσεων. Υπάρχει κάποια υπόθεση που τώρα εκδικάζεται και προβάλλεται πάρα πολύ και με την καταλάβετε πολιτικά. Η Γιούλεξ έχει μπλακεί. Μπορείτε να μα πείτε εσεί τι διεύθυνση μπορεί να υπάρξει, ούτω ώστε να μην ζημιωθεί και η Γιούλεξ και η αξιοπιστία τη Ένωση. Κρίμα γιατί αυτός που έρθει από το Κόσοβο αύριο ε, δεν θα είναι την ώρα που θα είμαι και εγώ εδώ για να τον ακούσω. Θα λείψω. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπράτνερ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σημεία στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία. Ε, όσον αφορά την πολιτική της ναυσιπλοείας βρήκα ενδιαφέροντα τα όσα είπατε, αλλά σε σχέση με την ε, Σομαλία, ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν συμπεριληφθήσαν στον προγραμματισμό. Ε, ακούγεται πολύ καλά το να ακούμε ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αλλά από όσο εγώ ξέρω, η Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού δεν συμπεριέλαβε συγγνώμη, τους εμπειρογνώμονες σε θέματα στρατηγικής ασφάλειας στην αυσιπλοεία στο σχεδιασμό της. Δηλαδή, στο επίπεδο θεωρίας τα πράγματα ακούγονται καλά, αλλά τελικά στην πράξη και στην εφαρμογή δεν είναι έτσι. Ένα άλλο ερώτημα όσον αφορά την ε, αυτοκριτική ε, σε σχέση με την πολιτικοστρατηγική συνεργασία στο Κονγκό. Ε, με εκπλήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναθεωρεί την εντολή της στο Κονγκό. Όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, ενώ εμείς κάνουμε σαν να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ε, βεβαίως ο στρατηγικός ε, παράγων είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια σχετική συζήτηση με ποιον εμείς μελλοντικά θα συνεργαστούμε στο επίπεδο της ε, μη στρατηγικής ε, παρέμβασης. Υπό, την έννοια, αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της στρατιωτικής στην πολιτική παρέμβαση και αντιστρόφως ε, νομίζω ότι δεν αξιολογούνται πολύ, ε, ε πάντοτε. Και πάντοτε όλα αυτά εξαγκράζουν στη θεωρία, αλλά είναι πολύ φτωχά στην πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θέλει να απαντήσει με το γύρο των απαντήσεων. Thank you very much for, uh, for all the questions. Uh, so see if we can structure them a bit. Uh, start with... Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Μα ε, έχει φύγει ο κύριος που έθεσε την ερώτηση. Και η κυρία Λόιζινγκ όμως έκανε την ίδια ερώτηση. Μίλησα για τον τοπικό πληθυσμό, είναι αμφίβολο για το, ποιος, το, το, το αν ενδιαφέρονται για το ποιος σας δίνει την περισσότερη βοήθεια. Φαντάζομαι πως αυτό σας εξαγρίωσε. Αναγνωρίζω όλες τις ευαισθησίες από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, από τις ΜΚΟ λοιπά για το στρατό, ε, αλλά εγώ μιλώ από την προοπτική του τοπικού πληθυσμού αυτή ήταν η, έτσι ίσχυε, ε, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα σχετικά έγγραφα, ότι το πρώτο που τους ενδιαφέρει δεν είναι ποιος τους δίνει τη βοήθεια. Και εντάξει, βέβαια υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα τρία. Το να δώσει κανείς βοήθεια σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό από την μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανοικοδόμηση. Αλλά για να απαντήσω και στον κύριο Φαν Μπάουερ, υπάρχουν φυσικά διάφοροι τομεί όπου ο στρατό χρειάζεται να έχει πόρου. Εγώ αναγνωρίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να εστιάσει την ασφάλεια. Να, δώσει, να παρέχει δηλαδή ένα ασφαλές ε, περιβάλλον, όπου δηλαδή οι ανθρωπιστικές οργανώσεις μπορούν να συνεργαστούν με τις πολιτικές αρχές και να μεριμνήσουν για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση. Θα πρέπει να βοηθήσουν και ε, τις ανθρωπιστικές ε, οργανώσεις ε, με όποια μέσο έχουν, αλλά με βάση τη ζήτηση, όχι με υποχρεωτική παροχή. Σε ορισμένε περιπτώσει, σε περιπτώσει δηλαδή που λείπει η ασφάλεια, πρέπει κανεί να γεμίσει το κενό. Αν δεν υπάρχουν δυνατότητε από τι αφγανικέ αρχέ, ή εν περιπτώσει από το χώρα υποδοχή, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια θα πρέπει ε, να μπορέσουν οι στρατιωτικές οργανώσεις, ο στρατό μάλλον να καλύψει αυτά τα κενά. Οι, οι κάτω χώρες έχουν μεγάλο ποσοστό αξιωματικών με πολιτικό ε, παρελθόν και στα σταδιοδρομία, νομικούς, μηχανικούς, εκπαιδευτικούς, προσωρινά μπορούν να στρατιωτικοποιηθούν και να προσπαθήσουν να καλύψουν αυτά τα κενά. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα σώματα γι' αυτό, ε, αλλά υπάρχουν και από άλλε χώρε ε, τέτοιοι ειδικοί και πιστεύω πως ο στρατός θα πρέπει να έχει τέτοιους πόρους στη διάθεσή του για να μπορεί να καλύπτει τα κενά Πολλοί κόσμος ε, επίσης ε, μιλά για τη σχέση μεταξύ της σταθερότητας, της ασφάλειας και της καλής διακυβέρνησης. Αλλά αν λειτουργεί κανείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που υπάρχει μεγάλη διαφθορά, όπου το Υπουργείο ε, Παιδείας δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει, είναι αγράμματο τελείως, αναλφάβητο, φαίνεται να είναι τρελό, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι από τις δυτικές πρωτεύουσες δεν καταλαβαίνουν πραγματικά ποια είναι η να γραψει ειναι αγραμματο τελειως αναλφαβητο φαινεται να ειναι τρελο αλλα πολλες φορες οι ανθρωποι απο τις δυτικε πρωτευουσες δεν καταλαβαινουν πραγματικα ποια ειναι η κατασταση Πολύ συχνά ακούμε δηλαδή ιστορίες ανθρώπων που έχουν πάει δύο μέρες εκεί και λένε ναι εγώ όταν πήγα στο Κονγκό και εννοούν ότι μείναν για δύο μέρες ε, είδα το Δίνα ή το Τάδε. Ε, καλή λοιπόν αξιολόγηση της τοπικής κατάστασης καταρχήν είναι πολύ βασική και έτσι μπορεί να φτάσει κανείς σε ένα άλλο συμπέρασμα ότι το στρατό χρειάζεται να έχει κάποιους πόρους για να μπορεί να γεμίσει αυτά τα κενά, να καλύψει αυτά τα κενά, εν πάση περιπτώσει να συνεργαστεί με τις αρχές, να δει ποιοι, ποιοι κάνουν τι, ποιοι είναι οι νομοθέτες, ποιοι έχουν την εξουσία. Και αυτό δεν είναι δουλειά στρατιωτική καθαρή. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ περισσότερη εναρμόνιση της ε, πολιτικής εμπειρογνωμοσύνης στα Υπουργεία Μήνης ή στις εξωτερικές συνεργασίες, ώστε να μπορούν δηλαδή οι στρατιωτικές μονάδες να καλύπτουν και τέτοιες ε, ανάγκες. Για τα όσα είπε η κυρία Σόνιγκ, ε, ε, ε, Λούνα Τσεκ, συμφωνώ πως πρέπει να δοθεί βάρος στο γυναικείο στοιχείο, γιατί μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση και να ενεργήσουν επ' Είδαμε θετικές αλλαγές για τη των τελευταίων χρόνων, δίνεται περισσότερη προσοχή, γίνεται πολλή έρευνα και στο ΝΑΤΟ αλλά και στους διάφορους στρατιωτικούς κύκλους Αλλά φυσικά είναι μία γυναίκα αξιωματικό σε 40-50. Αρκεί αυτό, δεν νομίζω αλλά υπάρχουν κάποιες θετικές αλλαγές. Και νομίζω πως έτσι απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Κρόιλ. Oui, euh, Madame euh, Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Έχετε απόλυτο δίκιο η κατάσταση στην οποία οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, δρούν και συγκεκριμένα ο Ερυθρό Σταυρό ε, δραστηριοποιείται, είναι όλα είναι και πιο επικίνδυνε. Και αυτό εδώ και αρκετά χρόνια. Λόγω του ότι. Στην ουσία αυτή η διαδικασία έχει επιταχυνθεί από το τέλος του ψυχρού πολέμου με ομάδες ε, αντίστασης ή αντιπολίτευσης που δεν έχουν πλέον τη στήριξη των διαφόρων μπλοκ και που αυτοχρηματοδοτούνται είτε προσφεύγοντας ε, παράνομα σε φυσικούς πόρους και το βλέπουμε αυτό πολύ καλά στην ε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είτε ενεργώντας με διάφορες άλλες μεθόδους, που παίρνουν κρατάνο μύρους και ούτω καθεξής και μάλιστα πολλές φορές δεν αναφέρονται καν στον αρχικό τους ε, ανώτερο. Αυτές οι ομάδες ε, μοιράζονται σε διάφορες άλλες ομάδες. Στην αρχή στον Ταρφούρ είχαμε δύο ομάδες επαναστατών και μετά πολλαπλασιάστηκαν. Πράγμα που σημαίνει βέβαια ότι οι επαφές γίνονται όλο και πιο δύσκολες και όπως το ξέρετε για να φτάσει κανείς από το σημείο Α στο σημείο Β μέσα σε μια κατάσταση ένοπλης σύραξης δεν φτάνουν τα εμβλήματα. Τα εμβλήματα εξαρτώνται από το πιο μέρος της σύγκρουσης έχουμε έρθει σε επαφή και αν αυτό το αναγνωρίζει. Τι κάνουμε λοιπόν, όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω, δεν έχουμε βέβαια θαυματουργές συνταγές, αλλά στην ουσία σεβόμενοι τις βασικές θεμελιώδεις αρχές, την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την οδετερότητα, γενικά μας αποδέχονται. Σε αυτή την υπόθεση το να μας αποδεχτούν είναι το βασικότερο στοιχείο. Πρέπει δηλαδή να πάσα στιγμή να επαληθεύουμε με κάθε μέρος εξήγηση ότι μας δέχονται, γιατί τη μια μέρα μπορεί να μας δέχονται και την επόμενη να δεχόμαστε απελητικές επιστολές. Άρα λοιπόν πρέπει κάθε φορά να ξαναεξηγούμε και να διευκρινίζουμε. Τώρα σε τεχνικό επίπεδο εμείς προσπαθούμε να καταρτήσουμε τους εκπροσώπους μας, τους απεσταλμένους μας, τους βάζουμε σε πραγματικές καταστάσεις όπου έχουμε συναδέλφους που παίζουν τους επαναστάτες, που κρατούν, ας πούμε, φτιάχνουν οδοφράγματα και που συμπεριφέρονται, εν περιπτώσει, αντιπαθητικά, ώστε οι απεσταλμένοι μας να μπορούν να αντιδράσουν, τους παρατηρούμε και μετά τους συμβουλεύουμε και τους διορθώνουμε. Φυσικά όλα αυτά δεν αρκούν. Ε, θέλει, πρέπει κανείς να περάσει από τη, ε, τη δοκιμασία επιτόπου και εκεί πρέπει να υπάρχει πειθαρχία σχεδόν θετική ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας και κάθε φορά ε, κάθε βράδυ δίνεται αναφορά για τις ε, μετακινήσεις. Και έπειτα και ένα τμήμα ασφάλειας ε, στη Γενέβη που συμβουλεύει τις αντιπροσωπείς και που συνδέεται άμεσα με τους διευθυντές των επιχειρήσεων. Δεν, είναι, δεν λαμβάνει αποφάσεις, δίνει τεχνικής φύσης συμβουλές, πώς να φτιάξει κανείς ένα μπούνκερ, πώς να ασφαλίσει μια, ένα κτίριο σε σχέση με δεχόμενους βομβαρδισμούς. Είναι μόνο τεχνική η μονάδα αυτή, δεν λαμβάνει αποφάσεις όπως ας πούμε στο ΝΟΙΕ που υπάρχει ένα τμήμα που αποφασίζει αν είσαστε στη φάση 1, 2, 3, 4 ή αντιστρόφως ανάλογα, εμείς έχουμε δώσει ευθύνη στον ε, αρχηγό της αποστολής που αλαμβάνει κάθε φορά την ευθύνη για την απόφασή του. Σας ευχαριστώ. Κύριε Έρχαρτ. Ναι. Αναφερθήκατε στην λειτουργία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά... ότι υπάρχουν εδώ πολλοί κίνδυνοι. Υπάρχουν ορισμένα κείμενα μελετητών ε, που αναφέρονται σε αυτό τον τρόπο λειτουργία των ανθρωπιστικών ομάδων νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο σφαιρική προσέγγιση. που είναι σε αντίθεση με την ε, που, θα, που θέτει το αίτημα να, να, σέβεται κανείς όλους τους ε, παράγοντες που λειτουργούν επί τόπου. είναι δύσκολο να, ή μάλλον λέω μιλής, είναι δύσκολο να ενταχθεί η μαλλον λεω με ειναι δυσκολο βοήθεια σε μια τέτοια είδους σφαιρική προσέγγιση. Εδώ υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι. Εμείς πολύ συχνά ε, τίνουμε να βλέπουμε την στρατιωτική συνεργασία σαν ένα θέμα τεχνικής φύσεως. Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδώσουμε την πλήρη πολιτική του σημασία ε, στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης πολιτικών στόχων, δηλαδή σε ένα στρατηγικό πλαίσιο και στην περίπτωση αυτή και από αυτή την προοπτική ε, θα πρέπει να πλαισιωθεί κατά τρόπο που είναι, να είναι καλό ε, για την ε, αποστολή. Και μία τελευταία παρατήρηση. Πολύ συχνά έχουμε λυπείς πληροφορίες από τη χώρα στην οποία μεταβαίνουμε. Ορισμένοι είπαν ότι οι στρατιωτικοί γνωρίζουν τι γίνεται στο Αφγανιστάν. Εγώ θα έλεγα όχι, δεν γνωρίζουν τι γίνεται στο Αφγανιστάν, γιατί ακριβώ δεν γνωρίζουν τον πολιτισμό τη χώρα. Ε, πολλοί Γερμανοί στρατιώτες ε, δεν γνώριζαν ακριβώς τι γίνεται εκεί, ε, ποια είναι η νοοτροπία των Αφγανών. Ε, γιατί έχουν άλλα πράγματα να κάνουν, θέλω να του επικρίνω, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όταν προγραμματίζουμε τέτοιου είδου δραστηριότητε, θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερε γνώσει που δεν μπορούν να αποκτηθούν παρά μόνο με την βοήθεια των τοπικών ε, παραγόντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράιτ. Νομίζω πολλές ε, ερωτήσεις απευθυνθήκαν σε εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους βουλευτές για όλες τις ερωτήσεις που μου απίφθηναν. Θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω αυτές όπως γνωρίζω. Καταρχήν, το, η ερώτηση για το Αφγανιστάν, του κ. Μπετικόφερ. Ε, το πρώτο σημείο που θα έπρεπε να θυμηθούμε εν σχέση με τις ε, αποστολές αυτές είναι ότι είναι στελεχωμένες κυρίως από συμβολές των χωρών, από συμφορές των χωρών μελών, ε, εισαγγελείς, ε, αξιωματούχους κλπ. σε εθελοντική βάση. Εναπόκειται στη δική τους κρίση κατά πόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Αυτό αφορά το μη στρατιωτικό σκέλος. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα για το στρατιωτικό σκέλος. Εδώ οι προκλήσει είναι πολύ μεγαλύτερες και ειδικά στο Αφγανιστάν για τους ε, λόγους που γνωρίζουμε όλοι μας. Ε, θα έλεγα και αυτό είναι ένα σημείο που ανέφερε, είπατε, ε, εκπρόσωπος κατά επανάληψη. Αντί να εστιάζουμε στον αριθμό του προσωπικού, είναι στο, στο επίπεδο της ποιότητας κατά πόσο υπάρχει προστιθέμενα αξία, κατά πόσο γινόμαστε αποδεκτοί από τον εγχώριο πληθυσμό ή από τις αρχές και, ή κατά πόσο συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά με το ΝΑΤΟ. Ε, ακούγοντας τον Γενικό Γραμματέα σήμερα, ε, είναι σημαντικό να δούμε τι σημασία δίνουμε στη UPOL η αποστολή εξτάζει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητε της, να τις παρατείνει ή να τις επεκτείνει μάλλον σε περισσότερες περιοχές του Αφγανιστάν εφόσον υπάρχουν υπαρκή πόροι. Εμείς από την Επιτροπή, και αυτό είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα συνεργασίας, θα εξετάσουμε κατά πόσο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες, ε, ε, ε, κάποια δημιουργία κατάρτισης αστυνομικών. Ε, ε, θα υπάρχει ένας ε, νέος επικεφαλής της αποστολής. Ο προηγούμενος σημείωσε πολλές επιτυχίες. Θα υπάρξουν κάποιες διαφορές. Νομίζω ότι θα ήταν εσφαλμένο να συνάγουμε από τον αριθμό του προσωπικού ότι η αποστολή δεν σημείωσε επιτυχία. Τώρα, Όσον αφορά τόσο είπε η κυρία Λούνα Τσακ για το Τσάντ, εγώ συμμετείχα με συναδέλφους από, το, από τη Γραμματεία του Συμβουλίου στον προγραμματισμό αυτή τη αποστολή. Και θέλω να σα υπενθυμίσω το εξή. Υπάρχουν 4-5 διαφορετικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συγκεντρωθούν ε, στη συνεκτίμηση αυτή τη αποστολή. Και θα ήθελα να αποτίσω τιμή στου συναδέλφου του στρατιωτικού προσωπικού που είχαν την πρωτοβουλία να επανέλαβαν να καλέσουν η Πετροπή να συμμετάχει ευθύ εξ αρχή στον προγραμματισμό. Και μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε διάφορε συνιστώσει, κάτι το οποίο είναι καλό αποτέλεσμα. Έχουμε τη στρατιωτική αποστολή αυτή καθ' αυτή, την ανθρωπιστική συνδρομή, ένα πρόγραμμα που οργάνωσε ο πρώην Επίτροπος Μισελ για την ε, ποροχή βοήθεια στα στρατόπεδα, ε, βοήθεια για την ε, κατάρτιση. Ε, ο αρχαιός επιτελείου ήταν Ιρλανδός κλπ. Είναι, ήταν σαφές ευθύς εξ αρχής ότι η αποστολή αυτή ήταν περιορισμένης διάρκειας και στη συνέχεια θα την αναλάμβαναν τα Ηνωμένα Έθνη. Ο πρώτος στόχος ήταν να παράσουμε σταθερότητα και ασφάλεια. Και εσείς οι ίδια είπατε ότι ίσως σώσαμε μερικές ζωές, αλλά συγγνώμη, δεν μπορεί κανείς να το λέει έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην υποτιμούμε τη σημασία του να σώσει κανείς ε, κάποιες ανθρώπινες ζωές. Επίσης είχαμε πολύ καλές ε, ε, σχέσεις με τις συνεργασίες με τους μη κυβερνητικού οργανισμούς. δεν θεωρώ ότι δεν ήταν αποτελεσματική προσπάθεια για να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση έστω σε μια περιορισμένη διάρκεια χρόνου. Δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτηση σας για το Κόσοβο. Ε, ε, δεν ξέρω. Ε, ίσως ο στρατηγός Ντουκαμόμ είναι πιο αρμόδιος να σας απαντήσει. Στο Κονγκό είχαμε δύο αποστολές, Σάκ και την Γιουπόλ. Και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα όπου μια από τις ε, αποστολές αυτές ε, συμμετέχει. Έχεις βίας σεξουαλικής στη χώρα και έχουμε αυτή την αποστολή η οποία ανάλογα με τις προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες βέβαια αυτών των ε, αποστολών, αλλά όλα αυτά δεν είναι σταθερά συνέχεια, μεταβάλλονται. Τώρα όσον αφορά την θαλάσσια ασφάλεια, αποφασίστηκε σήμερα στο Συμβούλιο να γίνει μια συνάντηση, να εξεταστούν οι εναλλακτικέ και να μπορέσουν στα πλαίσια της ΚΕΠΑ να αναπτύξουν και μια πολιτική για τη θάλασσα. Υπάρχει και μια έκθεση που είναι η συμβολή των στρατιωτικών. Πέντε ναύαρχοι γράψανε τη σχετική έκθεση που και αυτή εξετάστηκε στην συνάντηση με την EDA. ληφθεί υπόψη και από των στρατιωτικών. Αυτά έκανε όσον αφορά την ε, θαλάσσια επιτήρηση κομισιών και έτσι να υπάρξει τελικά κάτι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η πειρατεία βέβαια είναι μείζον θέμα. Ακριβώς και αυτό το αφορά η υπηρεσία που τώρα συγκροτείται η CMPT. Βεβαίω περιμένουμε να δούμε πώς θα, εξεταστεί, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Το Συμβούλιο βέβαια με επιφύλαξη εξετάζει το σύνολο των δεδομένων. Ποιο είναι, θα είναι το επόμενο βήμα. Αλλά πάντως υπάρχει η εμπειρογνωμοσύνη και υπάρχει και η σχετική ομάδα εργασία που βέβαια όλα αυτά είναι στοιχεία που θα μα βοηθήσουν ο πρόεδρο. Ευχαριστώ και νομίζω ότι τώρα ε, ακριβώ φτάσαμε στην ώρα που οφείλαμε να σταματήσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε όλου ε, όσου συμμετέσχουν. Ε, βέβαια θα μα απασχολεί αυτό μέχρι την επόμενη συνάντηση τη Υποπιτροπή για αυτό το θέμα, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο αφορά ε, όλο, όλο μας το, το, το φάσμα του έργου αύριο δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τον, ε, τον, τον ε, στρατηγό Λεμπόν. Nous nous retrouverons donc demain à h 9h et Τον στρατηγό Κερμαντών, λέει ο πρόεδρος, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων και κλεισμένο των θυρών όσον αφορά το, το, πώς θα υπάρξει αυτού του είδους ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, της ε, ΣΕΜ5 και, και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, ώστε να μπορέσουμε πάνω σε αυτό το θέμα να έχουμε μια ανταλλαγή απόψη. Είναι κάτι που δεν το έχουμε προετοιμάσει, ούτε το το